Αν ε, μου επιτρέπετε να σας ζητήσω να βάλετε τις κάρτες ε, στη σχισμή καταρχήν. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. And I close the... Λήξη. more less Πάνω κάτω λειτουργεί. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Αγαπητοί φίλοι, για τον κατάλογο ψηφοφοριών καταρχήν. Κανονισμός για την ιστορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κρισιάνης Κάριν είναι ο εισηγητής, πρόκειται για προσωρινή συμφωνία που επιτέχθη στον άτυπο τριμερή διάλογο. Άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. And I close the vote. Ευρεία υποστήριξη. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, δεν είναι μαζί μας. Το δεύτερο θέμα αφορά επίση την ιστορική αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή τη φορά έχουμε οδηγία. Πάλι εισηγητή, κύριο Κάριν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τεράστια υποστήριξη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα σκληρών διαπραγματεύσεων που εγκρίνονται από την Επιτροπή ΙΤΡΕ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημαντικό θέμα, ετοιμότητα αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια. Φλάβιο Ζωνονάτο είναι εισηγητή. Προσωρινή συμφωνία σε άτυπο τριμήρι διάλογο. Άρχεται ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Λήξη. Συγχαρητήρια στον και αυτή η πολύ σημαντική συμφωνία με πολύ μεγάλη υποστήριξη. Και περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Οργανισμός για τη Συνεργασία Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας Μόρτεν Χέλβεκ Πέτερσεν είναι ο εισηγητή. Ψηφίζουμε την προσωρινή συμφωνία που προέκυψε από τι διοργανικέ διαπραγματεύσει. Άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Λήξη. Και πάλι εδώ έχουμε ευρία υποστήριξη. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ και ολοκληρώνουμε την ψηφοφορία για σήμερα. Janusz. Janusz. How? Mr.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 Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σταματήσετε τις καυτές συζητήσεις. Σας ευχαριστώ. Επόμενο σημείο λοιπόν. Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας. Η συζητής είναι ο κύριος Σούλτσε. Και θα θέλαμε να εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης Έχουμε την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν υιοθετηθεί η πρόταση αυτή, θα θέσει τέλος ε, στην ε, αλλαγή ώρας που λαμβάνει η χώρα δύο φορές το έτος ε, σε κάθε κρατος μέλος, στα τέλη Μαρτίου και στα τέλη Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει ουσιαστικά προκαλέσει την προσοχή και του κοινού αλλά και των μέσων ενημέρωσης. Και τώρα θα συζητήσουμε στην Επιτροπή μας το θέμα αυτό. Θα ήθελα να καλέσω τον εισηγητή, τον κύριο Σούλτσα, να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ähm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά θέματα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά θεωρώ ότι και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό αν ακούσουμε τους πολίτες. Προσωπικά είμαι υπέρ της κατάργηση της αλλαγής ώρας ε, και είναι θετικό το ότι είχε υποβάλει μια τέτοια πρόταση η Κομισιόν και ανταποκρίθηκε έτσι αυτήν την πρωτοβουλία στο διαδίκτυο, οπότε η Ευρώπη μπορεί να κινηθεί και γρήγορα όταν θέλει. Βεβαίω όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνει δεν γίνονται τα πράγματα τόσο γρήγορα σε άλλες ε, περιπτώσεις, αλλά Τέλος να πω κάποια γενικά λόγια για τα προβλήματα και τις λύσεις. Αυτό το θέλουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, πάνω από 80% των ερωτηθέντων. Γνωρίζουμε επίσης ότι από οικονομική σκοπιά, π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας, εντάξει δεν είναι τόσο μεγάλες εφορέ όσο μας έλεγαν και όσο ήταν κάποτε. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες πτυχές. Ε, π.χ. πρέπει να δούμε ακριβώς τα ζητήματα βιομηχανικής ε, πολιτικής, ε, μεταξύ των οποίων στον τομέα της αεροπορίας υπάρχουν κάποια ζητήματα. Γνωρίζετε τις χρονοθυρίδες, τα σλότς τα οποία δίδονται, ειδικά με πτήσεις σε τρίτες χώρες. Θα μπορούσαν Ακριβώ να δημιουργηθούν προβλήματα εάν γίνει κάτι τέτοιο βραχυπρόθεσμα. Γιατί βεβαίω μπορεί να πηγαίνει ή να έρχεται ένα αεροπλάνο από μια χώρα όπου δεν αλλάζει η ώρα και να δοθεί δύο φορές ε, η ίδια χρονοθυρίδα. Αλλά ε, αυτό έγινε στην Τουρκία, επίσης καταργήθηκε η ώρα χωρίς ε, κανένα σοβαρό πρόβλημα η αλλαγή της ώρας. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που είναι κάπως πιο σημαντικά. Το ένα είναι το πώς θα γίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταργήσει την αλλαγή ώρας, αλλά τελικά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να πούν πώς θα γίνει αυτό, γιατί έχουμε χειμερινή ώρα και θερινή ώρα και πρέπει να συμφωνήσουμε μετά σε ποια ώρα θα μείνουμε. Και χρειαζόμαστε τους αναλόγους κανόνες γιατί δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει κανείς από το Άμστερνταμ στο Στρασβούργο και να διασχίζει το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, να φτάνει στην Γαλλία και στη χειρότερη των περιπτώσεων θα μπορούσε να αλλάζει τέσσερις φορές την ώρα. Δηλαδή να έχουν ημέν ε, θερινή και χειμερινή ώρα εναλλάξ. Ε, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να συμφωνήσουμε κάπου έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν το τι θα γίνει. Αυτό όμως είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Τα κράτη-μέλη δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια συνένεση. Γι' αυτό ε, δεν θα γίνει τον Απρίλιο φέτος η αλλαγή όπως είχε προτείνει η Κομισιόν και ο Ζαν Κλοντ Και προτείνω το εξής για την όλη αυτή υπόθεση. να καταργηθεί η αλλαγή της ώρας, ναι, αλλά από την προϋπόθεση ότι πριν θα συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό τα κράτη-μέλη για το πώς θα γίνει αυτό. Και εδώ πέρα θα θέλαμε να διατηρηθούν βεβαίως οι τρεις ε, ζώνες ώρας που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό συντονισμού, κάτι που είναι απόλυτος απαραίτητο. Αυτά δεν υπάρχουν και πάρα πολλά να πει κανείς. Εμείς ε, ως ιτρέ έχουμε μόνο μια γνωμοδότηση. Να πω κάτι για το πότε. Είπα δεν θα γίνει πρόθεσμα. Με τις έπαφες που είχα, με τη βιομηχανία, με την οικονομία, με πολίτες, με εκπροσώπους κομισιών, θα μπορούσε να γίνει τον Απρίλιο του 2020. Είναι κάπως φιλόδοξο, κάποιοι λένε ότι είναι και πολύ αργά. Αλλά ελπίζω να εκμεταλλευτώ τις επόμενες ημέρες για να το συζητήσουμε με τους κοιόδης εισηγητές. Δεν αναμένουμε και τεράστιες συζητήσεις. Κάποιοι θα καταλήξουμε για να κάνουμε την πρότασή μας. Αυτά από μένα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφε. Η κυρία Κούμπουλα τρέψω τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ε, γνωμοδότηση. Ο εισηγητής ε, τα είπε. Έχουμε μια καλή βάση εδώ πέρα προσωπικά με έχει απασχολεί το θέμα, το παρακολουθώ εδώ και καιρό. Η βιομηχανία, η έρευνα, τα ψηφιακά ζητήματα, η ενέργεια, όλα αυτά ε, δεν νομίζω να αποτελούν εμπόδιο ε, για το να μην γίνει η αλλαγή υπάρχουν και μετρήσεις ειδικά στον τομέα της ενέργειας ε, που δείχνουν ότι πια η εξοικονόμηση ενέργειας που γινόταν στο παρελθόν είναι ελάχιστη. Ζητήσαμε λοιπόν από την Κομισιόν να υποβάλει μια πρόταση και προσπάθησε η Κομισιόν να το κάνει γρήγορα. Εντάξει, τώρα Από ό,τι φαίνεται φέτος ε, το Μάρτιο θα αλλάξουμε την ώρα για τελευταία φορά. Αξί μπορεί να αναβληθεί. Η Κομισιόν πάντως έχει κάνει την ε, δικιά της δουλειά. Πρέπει και εμείς τώρα να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Ε, δεν νομίζω να σοκαριστούν και οι πολίτες. Στην αεροπορία είναι κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα θέλα να αναβληθεί για λίγο ακόμα η αλλαγή του συστήματος. Ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών επίσης είναι σημαντικός, γιατί μέχρι τώρα έχουν την επιλογή σε ποια ζώνη θέλουν να ανήκουν. Η Ισπανία έχει άλλη ζώνη από την Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη. Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να παραμείνει. Το σημαντικό είναι στην εσωτερική αγορά ε, να μην υπάρχουν παραπάνω από δύο ώρες ε, διαφορά μεταξύ δύο χωρών. Για να υπάρχει και μια συνοχή. Βεβαίω, εντάξει, υπάρχουν γεωγραφικές ε, πτυχές. Η Φιλανδία δεν έχει την ίδια ώρα με τη Σουηδία και την Γερμανία. Αλλά αυτό θα παραμείνει. Αλλά όχι παραπάνω από δύο ώρες διαφορά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κ. Καζνοντεύσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ από καιρού ασχολούμαι με το θέμα. Ασχολούμαι με το χρόνο φιλοσοφικά. Τον Χάιντεγκερ με τον Άγιο Αυγουστίνο που ασχολήθηκαν με το θέμα. Δεν ξέρουμε τι είναι ο χρόνος, φιλοσοφικά τώρα μιλώντας. Πάντα θεωρούσα ότι η αλλαγή της ώρας ήταν μια διοικητική πράξη, ε, λίγο βία και συμμερίζουμε την άποψη του εγώ πιστεύω αυτό που πιστεύει και μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μα, ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτή την αλλαγή τη ώρα. Δύο φορέ το χρόνο η αλλαγή τη ώρα με έναν αυθαίρετο τρόπο. Ε, οι μελέτε δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πιστικά επιχειρήματα για να συνεχιστεί αυτή η πρακτική. Αντίθετα, κάποιες μελέτες φαίνεται να δείχνουν ότι η αλλαγή της ώρας έχει αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. ήθελα να πω ότι δεν συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα. Υπάρχει ένα παράδοξο, βλέπετε. Ποιο είναι αυτό. Στη Μαδρίτη έχουν την ίδια ώρα όπως στην κεντρική Ευρώπη. Διότι δεν σέβονται το βιολογικό χρόνο. Υπάρχει ήδη μια διαφορά μεταξύ Βρυξελών και Βαρσοβίας, μια ώρα περίπου, όσον αφορά την ανατολή του ήλιου. Εγώ θα ήμουν περισσότερο υπέρ του να έχουμε εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη. Κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει σε ποια ε, ζώνη ε, χρονική θέλει να ανήκει. Να διατηρήσει την ώρα τη χειμερινή ή τη θερινή ή ό,τι άλλο θέλει. Αυτό πρέπει να αποφασιστεί μεταξύ χωρών. Συμφωνώ επίσης να παρατείνουμε λίγο τη συζήτηση είναι σημαντικό να υπάρχει ευρεία τοποθέτηση. Στην Πολωνία οι πολίτες θέλουν να τοποθετηθούν, να πούν αν προτιμούν τη χειμερινή ώρα ή τη θερινή ώρα. Ιδού. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την κυρίαρχη βούληση των πολιτών σε συνεργασία με γειτονικές βέβαια χώρες, με γειτονικές περιφέρειες διότι υπάρχουν οι συνέπειε που ήδη αναφέρατε. Ιδού λοιπόν, αυτά είχα να πω και σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που τοποθετηθήκατε, λέει ο Πρόεδρο, εν ονόματι της Άλτε. Ο κύριο Φέντερλ έχει το λόγο. Ευχ... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν είμαι σίγουρο ότι πολλοί από εμά που έχουμε εκλεγεί το 2014 θεωρούσαμε ότι το θέμα τη ώρα θα ήταν από τα σημαντικότερα ζητήματα για του πολίτε και δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα εργασιών της θεωρούσε ότι θα αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο θέμα και ότι θα εξεταστεί τόσο γρήγορα και ότι θα τύχανε τόσο μεγάλη υποστήριξη από τους πολίτες. Είμαι από αυτούς που κατέφθασα αργά σε αυτό το θέμα, το αναγνωρίζω. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα επί σειρά ετών, αλλά βλέπω ότι τελικά απέκτησε σημασία το θέμα και έχει αποκτήσει προτεραιότητα. Και φαίνεται ότι θέλουμε να σταματήσουμε αυτή την αλλαγή τη ώρα δύο φορέ το χρόνο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε καλή δουλειά. Η Ολλανδία, η Πολωνία και άλλα κράτη-μέλη, αρκετά κράτη-μέλη έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη αυτή την αλλαγή και είναι καλό ότι άκουσε αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ τον εισηγητή, έξοχη η εργασία του και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε τα εκρεμή προβλήματα με απλό τρόπο και βάσει συνένεση ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι καλό το ότι παρατείναμε την προθεσμία κατά ένα έτος και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να συνεχίσει την επεξεργασία του θέματος, νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα και μια περίοδο εφαρμογή ενό έτου είναι αρκετά καλή, όπω πρότεινε ο εισηγητή. Και όπως είπε και ο συγητής και πολλοί άλλοι, είναι σημαντικό να έχουμε μια καλή, ένα καλό συντονισμό για να μην καταλήξουμε σε ένα χάος. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια ε, θα επιτευχθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Όχι διότι έχουμε ιδεολογικέ δυνάμεις που καθοδηγούν το θέμα και συγκεκριμένα συμφέροντα, αλλά είναι απλώς θέμα ε, στήριξης των πολιτών. Οι πολίτε το ήθελαν και εισάκουσαν του πολίτε ε, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Επόμενο. Εκ μέρου των Πρασίνων. Σκλέτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Μπούζακ. Επί μακρόν τώρα, πριν μπω στο Κοινοβούλιο, παρακολουθούσα αυτό το πρόβλημα Άκουγα τι έλεγαν οι πολίτες και γνωρίζω ότι η έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δημόσια διαβούλευση έδειξαν ότι η πλειοψηφία των πολιτών θέλουν να παραμείνει η θερινή ώρα, διότι στην καθημερινή ζωή ε, αισθάνονται οι πολίτες ότι οι συνήθειές τους αλλάζουν να αλλάζει η ώρα και οι που ακολουθούν στην εργασία τους. Θέλουν να έχουν περισσότερες ώρες με το φως του ήλιου. Και ξέρουμε ότι για τη, η τεχνη, ο τεχνητό φωτισμός που χρησιμοποιούμε ακόμα και σε αυτή την αίθουσα δεν είναι πολύ καλός φωτισμός για την ανθρώπινη υγεία. Βλέπουμε ότι θερινή και χειμερινή ώρα, η αλλαγή της ώρας δημιουργεί προβλήματα υγείας. Υποστηρίζω την έκθεση. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταργήσουμε την αλλαγή της ώρας, τερινή και χειμερινή ώρα. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει φέτος. Το 2020 είναι μια καλή πρόταση. Εξελέγημεν από τους πολίτες και θα πρέπει να τους ακούσουμε. Αν θέλουμε να προωθήσουμε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στο εκλογικό μας σώμα. Θα πρέπει να δείξουμε με ένα απλό παράδειγμα ότι τους ακούμε τους πολίτες και τους λαμβάνουμε υπόψη στις ε, πολιτικές που διαμορφώνουμε. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για το όριο της χιλιετίας, όταν είχαν πει όλοι ότι θα σταματούσαν τα πάντα στον πλανήτη με την αλλαγή της χιλιετίας. Δεν θυμάμαι να διαβάσαμε στα ΜΜΕ ότι η ρωσική απόφαση για θερινή και χειμερινή ώρα ότι είχε κάποιες συνέπειες για τις αερομεταφορές. Για όλα αυτά τα αποτελέσματα, για τις δημόσιες διαβουλεύσεις, όταν όλα αυτά γίνονται, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η βιομηχανία έχει συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. 90% των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων φορέων υποστήριζαν την αλλαγή του συστήματος. Δηλαδή τελικά να έχουμε μόνο μία ώρα. Θερινή ή χειμερινή. Μία ώρα, χωρίς αλλαγή. Αγαπητέ συνάδελφοι, ευχαριστώ. Εκ μέρους της Γκουε, η κυρία Σακοράφα έχει το λόγο κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, νομοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο για την εποχική αλλαγή της ώρας θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1980. Ο στόχος της ήταν η εναρμόνιση των υφιστάμενων εθνικών πρακτικών και του προγραμματισμού για τη θερινή ώρα. Το Σεπτέμβριο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση οδηγία για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών τη ώρα με την αιτιολογία ότι πλέον αμφισβητείται από του πολίτε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορισμένα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα η πρόταση, ενώ επεσήμανε τη, συνα... τη σημασία της εναρμόνισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εύρυπνη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν προσδιορίσε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το εφιστάμενο νομικό καθεστώς, τα προβλήματα δηλαδή που επιχείρει να λύσει η νέα νομοθεσία. Άποψή μου είναι ότι η νέα πρόταση της Επιτροπής παρότι επικαλείται την απέτηση εκ μέρου των πολιτών, την προστασία τη υγεία και τη οδική ασφάλεια και την ανάγκη αποκατάσταση των τυχών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην εσωτερική αγορά, δεν παρέχει επαρκή τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα του τερματισμού των εποχικών αλλαγών τη ώρα. Ειδικότερα λοιπόν θέλω να επισημάνω ω προ το θέμα τη αμφισβήτηση εκ μέρου των πολιτών του φυστάμενου καθεστώτο. Θεωρώ ότι η δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε δεν ήταν αντιπροσωπευτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω προ το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο του 2018. Η πρόταση τη Επιτροπής δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση τη φυστάμενη νομοθεσία οδηγία, όπω ρητό ζητήθηκε και ω εκ τούτου παραμένει υπό αμφισβήτηση η ανάγκη αναθεώρησή τη. Ω προ τι εθνικέ θέσει. δεν βλέπω να υπάρχει συμφωνία. Γνωρίζω ότι σχεδόν ομόφωνα τα κράτη μέλη απέρριψαν την πρόταση της Αυστριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών το Δεκέμβριο. Η συντριπτική του λοιπόν πλειοψηφία έχει εκφράσει την ανάγκη για προηγούμενη διαβούλευση με του αρμόδιου φορεί και του πολίτε, την ανάγκη για τον έλεγχο των συνεπειών τη επιλογή μόνιμη θερινή ή χειμερινή ώρα σε όλου του τομεί και ιδίω του κόστου που θα προκαλέσει, την ανάγκη συντονισμού μεταξύ των γειτονικών κρατών μελών για την επιλογή μόνιμη ώρα ω προ την αποφυγή δημιουργία παραπέρα προβλημάτων και κυρίω την ανάγκη να καταστεί σαφή ο λόγο για τον οποίο τα κράτη-μέλη καλούνται να αποφασίσουν τη μετάβαση από ένα σύστημα εναρμονισμένο και ρυθμισμένο εδώ και χρόνια σε ένα άλλο, το οποίο απορριθμίζει μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση με προφανείς τις δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πράγματι, από το σκοπό και το περιεχόμενο της πρότασης διαπιστώνεται ότι δεν στοχεύει στη δημιουργία ενός εναρμονισμένου καθεστώτος για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αντίθετα, τίθεται μόνο η υποχρέωση τη κατάργηση των εποχικών αλλαγών τη ώρα. Ενώ εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, όπω είπα και προηγουμένω, να επιλέξουν την ώρα που επιθυμούν σε μόνιμη βάση. Πρόκειται ακριβώ για αυτή την έλλειψη εναρμόνιση που θα δημιουργήσει διαφορετικέ καταστάσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα λειτουργήσει αρνητικά στην εσωτερική αγορά. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταλήγοντα, θέλω να υπογραμμίσω. Αν το θέμα μα σήμερα είναι η κατάργηση τη νομοθεσία, η οποία έχει επιφέρει προβλήματα στην υγεία των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οδική ασφάλεια, δεν θα συζητούσαμε παραπέρα τα αυτονόητα και θα αποφασίζαμε όλοι ομόφωνα να θεσπίσουμε μια νέα νομοθεσία για την προστασία των πολιτών το συντομότερο δυνατό. Με δεδομένο όμω ότι ο κύριο σκοπό τη οδηγία ήταν και παραμένει η εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και ιδιαίτερα η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τομέα των μεταφορών, θα πρέπει να σκεφτούμε εκ νέου τις συνέπειες της απορρίθμιση που επιχειρείται με την πρόταση αυτή, καθώς και το κόστος που θα επιφέρει στα κράτη-μέλη. Υπό το φως λοιπόν όσον ανέφερα προηγουμένως, θεωρώ απολύτως απαραίτητο η Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη επιπτώσεων και να τεκμηριώσει πλήρως τους λόγους για την αναγκαιότητα αυτής της σημαντικής αλλαγής που επιχειρείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η πρόταση οδηγίας γίνει αποδεκτή υπό την ήδη υπάρχουσα μορφή τη. είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που πιστεύουμε ότι επιχειρεί να λύσει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές. Ο κύριος Βέρνερ Λάγκεν είναι ο πρώτος που έχει ζητήσει το λόγο. Pardon, pardon. Συγγνώμη, συζητούσα με τον εισηγητή. Ε, Θέλω να εκφράσω και εγώ την ε, άποψή μου και να συμφωνήσω με την τελευταία ομιλήτρια της ΓΚΟΕ. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ανώριμη. Καταστρέφει την εσωτερική αγορά, τα αφήνει όλα στα κράτη-μέλη και δεν ξεκαθαρίζει το θέμα ζώνη ώρας και αλλαγή της ώρας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν την ώρα. Αυτό είναι ε, εθνικό δίκαιο. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για την εσωτερική αγορά. Λοιπόν, αν περάσουμε εμείς αυτή την πρόταση, εντάξει μπορεί να υπερψηφιστεί, εγώ θα καταψηφίσω. Αλλά ε, το επιχείρημα πριν από τον προηγούμενο αιώνα όταν άλλαξε η ώρα ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας. Πράγματι εντάξει μπορεί να μην είναι τόσο πολύ θέμα. Τώρα μας λένε για την υγεία των ανθρώπων. Ε, μπορούμε να δούμε λοιπόν, ε, αλλά κοιτάξτε, μιλάτε για 4,2 εκατομμύρια ερωτηθέντες, 3 εκατομμύρια ήταν από τη Γερμανία οι περισσότεροι ήταν κατά. Και θέλανε, τι θέλανε αυτοί, μόνιμη θερινή ώρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θέλαν να αλλάξουν κατ' ουσίαν ζώνη ώρα. Και ξαφνικά γίνεται προτεραιότητα τη Κομισιόν. Όχι, δεν είναι. Οι λόγοι κατά της αλλαγή είναι πολυεπίπεδοι και σημαντική. Και καλά θα κάνει το Κοινοβούλιο να κάνει μια μελέτη επιπτώσεων. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι για το ότι έχουμε ακόμα 26 ε, μέρες μέχρι την επόμενη αλλαγή ώρα. Σας ευχαριστώ. Όχι, 62, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήμουν ε, κατά των αλλαγών όλη μου τη ζωή όταν εξελαγή στο Ευρωπαϊκό Γενοβουλίο πριν 10 χρόνια. Συνειδητοποίησα ότι ε, ασχολούμαστε με το θέμα υπό την προεδρία του Χέρμπεν Γάιλ και χρειαστήκαμε 7 χρόνια για να πείσουμε την Κομισιό να κινηθεί επί του θέματος και έχουμε μόνο ω απάντηση στη δημοσιογραφική βούλευση μπορεί να προωθήσει η Κομισιόν την πρόταση. Έτσι λοιπόν, αν ε, θέσουμε τέλο στην αλλαγή τη ώρα, αυτό θα είναι μεγάλη νίκη για το Κοινοβούλιο. Θα δείξουμε ότι λειτουργεί το Κοινοβούλιο και ότι οι πολίτες έχουν εξουσία και μπορούν να κινητοποιήσουν την Κομισιόν. Τώρα, στη δημόσια διαβούλευση πάνω από το 80% όσων απάντησαν ε, ήθελαν να τεθεί τέλος στην αλλαγή της ώρας και και οι περισσότεροι από αυτούς ε, ήθελαν τη θερινή ώρα μας ε, ξέπληξε βέβαια και μας χαροποίησε ε, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, ανέφερε στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ότι θα γινόταν η αλλαγή αυτή το 2019. Το 2019 μάλλον είναι πολύ νωρίς, το 2020 έχει νόημα για μένα και τώρα εξετάζουν οι χώρες τι θα κάνουν. Και στην Ιρλανδία υλοποιούμε και εμείς δημόσια διαβούλευση για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά βέβαια από τους ανθρώπους που συναντώ στο δρόμο η ευρεία πλειοψηφία θέλει να τεθεί τέλος σε αυτή την ε, αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο και νομίζω ότι έχουμε την υποχρέωση να ακολουθήσουμε τη βούληση των πολιτών. Τώρα, ίσως ε, κάποια χώρα να κρατήσει τη χειμερινή ώρα και κάποια άλλη χώρα τη θερινή ώρα. Ε, όμως ε, είναι καλύτερο από το να αλλάζουμε την ώρα δύο φορές το χρόνο και θυμάμαι ότι οι ΗΠΑ ε, έχουν διαφορετικές ζώνες και όλο το χρόνο και μιλάμε για μία χώρα. Έτσι λοιπόν δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να σταματήσουμε την βούληση των ανθρώπων να εφαρμοστεί ε, αυτή η πάυση της γελίας ε, πρακτικής ε, του να αλλάζουμε την ώρα δύο φορές το χρόνο. Ε, νομίζω ότι και ο Μπέρναρ Λάγκιν θα μπορούσε να μας πει και δύο λόγια για τη βούληση του πρώην συναδέλφου που θα μας αφήσει αυτή την ωραία κληρονομιά αν εθετήσουμε την πρόταση. Ευχαριστώ, κύριος Μπλάνκο. Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα συζητούμε την αλλαγή της ώρας, μία από τις αποφάσεις που έχουν ορατό και άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Όμως η αλλαγή της ώρας δεν μπορεί να γίνει ελαφρά την καρδία καθώς έχει διάφορες επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις, ενεργειακές επιπτώσεις, την ασφάλεια της κυκλοφορίας αλλά και στις συνήθειες και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί πολλάκις επί του θέματος. Η τελευταία φορά ήταν πέρσι όταν ε, απευθυνά έκκληση στην Κομισιόν να κάνει μια εξαντλητική αξιολόγηση της οδηγίας 2084 ε, και να παρουσιάσει, αν είναι απαραίτητο, μια πρόταση για την αναθεώρησή της. Έτσι, λοιπόν, ζητήθηκε εξαντλητική αξιολόγηση και λυπάμαι, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Επίσης, αν και ξέρουμε ότι υπήρχε αυτή η δημόσια διαβούλευση και είχαμε πάρα πολύ υψηλή συμμετοχή των πολιτών, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 70% οι απαντήσει προέρχονται από τη Γερμανία. Οι πολίτε που απάντησαν είναι από τη Γερμανία κατά 70%. Έτσι λοιπόν αυτό το θέμα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Το 70% των απαντήσεων προέρχονται από τη Γερμανία. Επομένω, δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιπροσωπευτικότητα του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να αμφισβητήσουμε τη διαβούλευση. Επομένως, ο κίνδυνος που διατρέχουμε σήμερα είναι ότι αν βιαστούμε, χωρίς να έχουμε την μελέτη αντικτύπου, να καταλήξουμε να λάβουμε αποφάσεις που δεν θα έχουν βάση και δεν θα αιτιολογούνται και έτσι θα δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα και θα δημιουργήσουμε σύνορα εκεί που δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, εγώ δεν κρίνω αυτή τη στιγμή την απόφαση, αλλά πριν να προχωρήσουμε θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και επιτακτικό να αναλύσουμε εις βάθος τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η απόφαση και έτσι έχει ζητηθεί και από αυτό το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφο. Η κυρία Γκροστέτη, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ειλικρινά, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θεωρώ ότι κάπως επιπόλαια χειρίζεται το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με κάποιους συναδέλφους που μόλις είπαν ότι η μελέτη αντικτύπου δεν υπάρχει στην πραγματικότητα και δεν έχουμε εξετάσει όλες τις συνέπειες αυτής της αλλαγής της ώρας. Εγώ άκουσα έναν από του συναδέλφου που εκτιμώ πολύ, αλλά μα είπε ότι τελικά τοποθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι πολίτε. 4,5 ε, εκατομμύρια πολίτε ε, στα 600 εκατομμύρια στην Ευρώπη, τι σημαίνει. Και είναι αλήθεια ότι η ευρία πλειοψηφία των απαντήσεων προέρχεται από τη Γερμανία. Επομένω, ε, αυτό δεν είναι ενδεικτικό δεν ε, ρωτήσαμε τους ε, πολίτες ε, στις βόρειες χώρες, στις χώρες ανατολικά ή στις χώρες του Νότου. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα γιατί αυτό το θέμα είναι εθνική αρμοδιότητα. Όμω, αν ο καθένα αποφασίσει τι θέλει στη δική του γωνιά, θα είναι καταστροφικό το αποτέλεσμα και θα είναι κατά τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, λοιπόν, εγώ στην περίπτωση αυτή είμαι εντελώ αντίθετη σε μια τέτοια απόφαση η οποία δεν θα εξυπηρετήσει την εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και σκεφτείτε τι γίνεται και με του εποχικού εργαζομένου. Έχουμε πολλού Γάλλους που εργάζονται στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Φανταστείτε να μην είναι το ίδιο το ωράριο στις χώρες αυτές. Φανταστείτε τι καθημερινέ επιπλοκές που θα έχουν οι εποχικοί εργαζόμενοι. Έτσι λοιπόν, α μελετήσουμε ει βάθο τα πράγματα πριν να λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορλίτσεκ, παρακαλώ. Επόμενος ομιλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπαν, νομίζω, οι προλαλήσαντες. Είτε θα έπρεπε να κάνει μια ουσιαστική ανάλυση η Κομισιόν, ή να πει ότι εμείς θέλουμε να καταργήσουμε την αλλαγή της ε, ώρας και να συμφωνήσουν μετά στο Συμβούλιο τα κράτη, να συμφωνήσουν όμως πώς θα έπρεπε να το κάνουν. Αλλά εδώ πέρα πραγματικά ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο είναι ξεκάθαρο απλό και το οποίο δεν έχει πραγματική βάση η αλλαγή της ώρας. Ε, όταν εισήχθη είχε κάποιο νόημα, είχε κάποια επιρροή, είχε και κάποια βάση στο θέμα της ενέργειας. Ε, σήμερα δεν έχει πια νόημα. Και το επιβεβαιώνω πράγματι ότι είχε κάποια σημασία στα αργοστάσια τότε. Αυτό το οποίο είπε τώρα ο κύριος Λάγκεν και η κυρία Σακοράφα έχουν απολύτως δίκιο. Και πράγματι και εγώ θα ήθελα να το αφήσουμε στα εθνικά κράτη. Ε, δηλαδή να πούμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να καταργηθεί η αλλαγή της ώρας και να το αποφασίσει μετά το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ, κυρία Βίρκουνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σχέδιο γνωμοδοτήσεω του εισηγητού. Αντιπροσωπεύω του Φιλανδού πολίτε και πρέπει να πω ότι στη Φιλανδία οι πολίτε ήταν πολύ κατά τη αλλαγή της ώρας κάθε χρόνο και πέρσι στην πρωτοβουλία των πολιτών αυτή πέρασε από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο, είχε μεγάλη υποστήριξη και η κυβέρνηση Φιλανδίας θέλει να αλλάξει αυτή την οδηγία. Ξέρουμε ότι είναι πολύ παλιωμοδίτικη η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο. Στην αρχή η ιδέα ήταν εξοικονόμηση ενέργειας, τώρα ξέρουμε ότι η τεχνολογία είναι πολύ καλύτερη τώρα και δεν έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Νομίζω επίσης ότι στην Επιτροπή Ήτρε πρέπει να εστιαστούμε επί της βιομηχανίας και του ενεργειακού τομέα και τι είδου ωφέλη αποκομίζουν από την αλλαγή της ώρας φορέ στον χρόνο και ξέρουμε ότι δεν αποκομίζουν ωφέλη, περισσότερο επιβλαβήν τα αποτελέσματα. Είναι πολύ καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να σταματήσουμε αυτή την πρακτική, την εφαρμογή τη οδηγία και εγώ θα έλεγα ότι εξεπλάγει και χάρηκα ιδιαίτερα διότι δραστηριοποιήθηκε τόσο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο ξέρουμε ότι η συζήτηση την διεξάγουμε επί σειρά ετών και στα κράτη-μέλη και ζητούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποια πρόταση. Μετά από τη δημόσια διαβούλευση, είπαμε, και νομίζω ότι δραστηριοποιήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα στην Κομισιόν και χάρη καλώ ιδιαίτερω. Και νομίζω ότι δεν είναι πολύ δίκαιο τώρα να λέμε ότι μόνο οι Γερμανοί συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση, ότι ξέρουμε ότι σε πάρα πολλέ χώρε οι πολίτε ήταν πάρα πολύ ενεργοί και συμμετείχαν, αλλά υπήρχαν διαφορέ σε κάποιε χώρε δεν είναι το σημαντικό θέμα, σε κάποιες άλλες χώρες όμως είναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν τώρα το ότι προχωράμε α, όσον αφορά αυτή την πρόταση, αλλά νομίζω ότι το μεγάλο σφάλμα ήταν ότι δεν είχαμε συντονισμό, επαρκή συντονισμό στην αρχή, διότι σε πολλές χώρες τώρα γίνεται συζήτηση αν θα πρέπει να επιλέξουν θερινή ώρα, χειμερινή ώρα και περισσότερο συντονισμό απαιτείται τώρα, διότι έχουμε διαφορετικές ζώνες ώρας στην Ευρώπη, άρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για συζήτηση, διότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίση να συζητήσουν μεταξύ του ε, ποια... και να συζητήσουν και εντό των χωρών ποια ώρα θα επιλέξουν. Αλλά η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μάισνερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω και εγώ με την κυρία Βιρκούνεν, ε, συμφωνώ με την Κομισιόν και τον κύριο Σούλτσε και τον κύριο Πράγματι, όταν εισήχθη αυτό το σύστημα, σκεφτόταν ότι θα εξοικονομήσουν ενέργεια. Εν τω μεταξύ δεν ισχύει, εξοικονομούμε ενέργεια το καλοκαίρι, το βράδυ, αλλά ξοδεύουμε περισσότερη ενέργεια το πρωί. Υπάρχει κόσμος που έχει ηλιακά πάνελ και παρόλα αυτά το πρωί ανοίγει τη θέρμανση γιατί δεν έχει βγει ο ήλιος. Οπότε ε, το τελικό αποτέλεσμα είναι μηδέν. Και γίνονται ατυχήματα. Μα θέλω να μιλήσω. Ε, το πρωί με τα παιδιά που πάνε σχολείο επίσης. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να το καταργήσουμε. Ε, αν ο στόχος έχει επιτευχθεί, πρέπει να καταργήσουμε την ομοθεσία. Υπήρχε ο στόχος αυτό, ο στόχο αυτό επετεύχθη, Τελείως, Υπάρχουν και άλλε χώρε. Και η Ρωσία το έχει κάνει. Είδε, δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό το κατήργησαν. Και βιολόγοι, ε, νομπελίστες έχουν παρατηρήσει ότι άνθρωποι και ζώα προσανατολίζονται με βάση τα άστρα και το φυσιολογικό είναι να μην υπάρχει αλλαγή ώρας. Ε, και μας είπανε ότι το λογικότερο θα ήταν η χειμερινή ώρα. Τώρα εντάξει, αυτό είναι θέμα απόφασης ε, αν θα είναι η χειμερινή ή θερινή. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά αποδεδειγμένα ένα ποσοστό 20% των Ευρωπαίων, η ε, χρόνια άρρωστοι, τα παιδιά οι ηλικιωμένοι, αποδεδειγμένα δηλαδή στην αλλαγή της ώρας και αμέσως μετά εκδηλώνονται πολύ περισσότερες ε, ασθένειες και πέφτει η συγκέντρωση των παιδιών, πέφτουν οι βαθμοί τους στο σχολείο. Αυτά φαίνονται. Εντάξει, μετά αποκαθίσταται, αλλά ε, δεν πρέπει να. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα. Και βεβαίω, εντάξει, ναι, τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα, πάντα έτσι ήταν. Γιατί θα αποφασίσουν ε, το τι θέλουν. Και επειδή θέλουν την εσωτερική αγορά, ε, συμφώνησαν πράγματι σε μια ώρα και στην Ελβετία. όταν είχε γίνει η αλλαγή της ώρας έγινε δημοψήφισμα στην ε, Ελβετία. Ο πληθυσμό ήταν κατά. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση είπε ότι θα ακολουθήσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν μπορούμε να έχουμε άλλη ώρα από τι γειτονικέ χώρε. Ε, λοιπόν, αυτό είναι και ένα επιχείρημα ε, όταν μιλάμε για την κοινή αγορά και επίσης αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στα δρομολόγια, στις μεταφορές κτλ. Καλό είναι να έχουμε μία ώρα μονίμως. Γνωρίζω τέλος ε, το είχα συζητήσει με τον Επίτροπο Κάλλας ε, πριν από δύο χρόνια και μας είπαν εντάξει φοβόμαστε ότι θα δημιουργηθεί ένα μοσαϊκό όπως λένε οι συνάδελφοι. Ε, βασίζομαι στη λογική των κυβερνήσεων ότι θα λειτουργήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ καυτό θέμα. Έχω και άλλα καινούργια ονόματα μιλήτων στον κατάλογο, μακροσκελέστατος κατάλογος συναδέλφων που θέλουν να μιλήσουν. Επόμενος. Η κυρία Γκρίφιν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Ζέρζη. Απαντώντας στα σχόλιά σου θα είμαι σύντομη. Να υπογραμμίσω κάτι. Βέβαια για την Επιτροπή μας θέλουμε να δούμε τον αντίκτυπο για τη βιομηχανία που έχει αλλαγή της ώρας. Ποιος είναι ο οικονομικός αντίκτυπος. Αλλά όπως είπε μόλις τώρα ο συνάδελφος, η συνάδελφος πρέπει να δούμε και τις συνέπειες στην υγεία. Σαν Ήτρε όλο το χρόνο είχαμε προσέγγιση βιομηχανικής. Βιομηχανική, αλλά θέλαμε να δούμε βιομηχανικές ε, συνέπειες, κοινωνικές συνέπειες και αντίκτυπο στην υγεία. Ε, έχουμε πολλές στοιχείες να εξετάσουμε, πολλή δουλειά ακόμα να γίνει όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταμπουράνο είναι επόμενος και εγώ θα είμαι σύντομο, διότι πολλοί θέλουμε να μιλήσουμε. Πιστεύω ότι χρειάζεται μελέτη αντιχτύπου ευρέω φάσματο, να δούμε τι γίνεται από πλευρά ιατρική, ε, βιολογική, ε, στην εσωτερική αγορά και τη βιομηχανία. Δεν σοφό να πάρουμε μια απόφαση χωρί να γίνει αυτή η μελέτη. Και πιστεύω ότι να αφήσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν το σύστημα ή όχι δεν είναι ούτε αυτό σοφό, διότι θα οδηγούσε σε άλλα προβλήματα όσον αφορά το εσωτερικό εμπόριο, επικοινωνίες, συναλλαγές και τη συνεργασία παραγωγική μεταξύ των κρατών ε, μελών. Αυτά και σταματάω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Μαρτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν, θα είμαι σύντομος. Αλλά αυτό που κατανοώ από τη συζήτηση ότι πρέπει να περιμένουμε όχι δεκαετίες, αλλά είναι επίγον να πάρουμε το χρόνο και να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Και θεωρώ ότι είναι κάπως ε, βιασμένο, κάπως είναι θρασί από την πλευρά της Κομισιόν ε, να βασίζεται σε αυτή τη ε, διαβούλευση. Γιατί τελικά χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά η Κομισιόν, ανάλογα με τα συμφέροντά της. Εγώ συμφωνώ με όσα προτάθηκαν για τη μελέτη αντικτύπου και ακόμη και αν πρόκειται για αρμοδιότητα των κρατών μελών, θα πρέπει τα κράτη-μέλη στην περίπτωση αυτή για να μπορούν να έχουν την πιο την πιο ευρεία εικόνα, να υπάρξει διαβούλευση σε κάθε κράτο μέλο για να δούμε αν οι πολίτε συμφωνούν ή όχι για την αλλαγή τη ώρα. Και κατόπιν θα συζητήσουμε και θα δούμε ποια ζώνη ώρα θα υιοθετήσουμε, τη χειμερινή ή τη θερινή, γιατί ο καθένα, αν κρατήσει την ώρα που θέλει, δεν σα λέω τι χαμό θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν, γιατί το θέμα αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και πολιτικό και είναι πολύ σημαντικό και για τις μελλοντικέ ευρωεκλογέ. Όλοι μας θα ρωτηθούμε γιατί μέσα σε δέκα χρόνια η Κομισιόν ε, δεν έχει αναλάβει καμία δράση, το χάρη στο να θέσει τέλος την αλλαγή της ώρας. Δεν είναι λοιπόν απλώς οικονομικό το θέμα. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα και οικονομικό και, και οικονομικά και πολιτικά. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να μας παρουσιάσει τις προτάσεις της το συντομότερο. Θα πρέπει να μας παρουσιάσει Μα αν, αν μα παρουσιάσει μια μελέτη εκδικτική, που δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό τίποτα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ, όπω είπε ο κ. Λάνγκεν, θα πρέπει να αποφασίσουμε βάσει τη περιφερειακή ε, αρχή. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε την εξή κατάσταση, να έχουμε άλλη ώρα στη Λιθουανία και στη Λετωνία 200 χιλιόμετρα μακριά να έχουμε άλλο ωράριο όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να έχουμε την ε, απαραίτητη εξουσία για να αλλάξουμε την ε, απόφαση και να εφαρμόσουμε κάτι έτσι ώστε να μην αλλάζει συνεχώς η ώρα. Ναι. Σας είχα στον καταλογό μου, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Απλώς ήθελα να αποσαφηνίσω, γιατί άκουγα διάφορες μεταφράσεις και εγώ έχω την ίδια με τον κύριο Καρσανεύσκη δεν εννοούσα ότι θα πρέπει να έχουμε τρεις διαφορετικές ε, ζώνες ε, ώρας ε, στα διάφορα κρατημέλια, αλλά μέσα στο διακρατισμό δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικές ώρες. Και εξεπλάγει που είπαν κάποιοι ομιλητές, ε, αναφέρθηκαν στις ζώνες ε, ώρας. Δεν υπάρχει σήμερα συντονισμός. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν όποια ζώνη ώρας θέλουν. Η οδηγία αυτή δηλαδή δεν αλλάζει αυτό το συντονισμό. Αλλάζει μόνο το εξής, ότι δεν θα περάσουμε από τη θερινή ώρα στη χειμερινή ώρα και δεν θα αλλάζουμε δύο φορές το χρόνο την ώρα. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω τώρα είναι πολιτική, είναι παρεξήγηση, πάντως ε, δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε ε, τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ να περιοριζόμαστε στα γεγονότα όταν νομοθετούμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα είναι πολύ εύκολο να αποφασίσουμε τα πάντα μεταξύ των κρατών μελών. Ε, δεν θα είναι εύκολο, είμαι σίγουρος. Γιατί θέλουμε να λάβουμε υπόψη και την άποψη των πολιτών. Και η άποψη των πολιτών θα μπορούσε να διαφέρει στα κράτη-μέλη που μπορεί να βρίσκονται και πολύ κοντά το στο άλλο. Δεν είναι εύκολο λοιπόν, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Εφόσον ξεκίνησαμε αυτήν την ιδέα, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Και εγώ γενικά έχω κάποιε αμφιβολίε, αλλά νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να προβούμε σε ένα σωστό έλεγχο και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Μπορούμε λοιπόν να, υποστηρίξουμε την δεύτερη με πλήρη ενθουσιασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σήμερα από τον κύριο Ντεμάγερ από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΟΥΒ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Γιώργεν για αυτήν την τζιμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Σούλτσε, για το σχέδιο γνωμοδότηση και την Επιτροπή για την στήριξή τη αναμένουμε και την τελική σας γνωμοδότηση εν καιρό αναγνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί λίγος ε, χρόνος ε, για να εφαρμοστεί λίγος περισσότερος από ό,τι είχαμε προβλέψει στην πρότασή μας και αναγνωρίζουμε επίσης ε, την ανάγκη για μια συντονισμένη προσέγγιση για να γίνει αυτό με έναν τρόπο επιτυχή για τους Ευρωπαίους πολίτες αναγνωρίζοντας πλήρως όπως υπόθηκε ότι η επιλογή της ζώνης ώρας είναι εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών και γνωρίζουμε ότι πολλά κράτη-μέλη κάνουν αυτή τη στιγμή την εθνική διαβούλευση και αξιολόγηση για να καταλήξουν σε μια επιλογή ε, ζώνης ώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, ο συνάδελφος ο κ. Μπαλτσίτης. Ναι, ναι, ε, είναι επίμαχο το θέμα. Ε, γίνει και δεύτερος γύρος συζήτησης. Ο κ. Μπλάνκο Λόπες. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Απλώς να κάνω μια διευκρίνηση. Νομίζω ότι δεν είναι σκόπιμο ούτε κατάλληλο εκπρόσωπος της Κομισιόν να λέει ότι ικανοποιήθηκε που η πλειοψηφία της Επιτροπής αυτής ε, ήταν υπέρ της πρότασης της Κομισιόν, γιατί ακόμη δεν έχουμε ψηφίσει για το θέμα αυτό και αν άκουσα καλά, εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι ομιλητές αμφισβήτησαν το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν ε, είχε κάνει μελέτη αντικτύπου πριν να παρουσιάσει την πρωτοβουλία. Τουλάχιστον εγώ αυτά κατανόησα. Uh, uh, well, we've got some doubts. Κοιτάξτε, έχουμε κάποιες αμφιβολίες, αλλά σε γενικές γραμμές στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιες επιφυλάξεις και υπογραμμίσαμε πολλές επιφυλάξεις στην συζήτησή μας. Το γνωρίζουμε. Λοιπόν, ο κ. Λάγκεν, ξανά μια ερώτηση. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Η ερώτησή μου είναι, η αξιολόγηση αντικτύπου τι γίνεται, την έχετε αναθέσει, την κάνετε ή απλά αγνοήσατε αυτό το οποίο σας ζήτησε το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Εγώ αναφέρθηκα στο ότι χρειάζεται χρόνος για να συμφωνηθεί και να εφαρμοστεί γιατί προέβλεπε η πρόταση της Κομισιόν ότι θα σταματούσε τώρα η αλλαγή της ώρας δηλαδή από την επόμενη φορά και αναγνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Ε, στην πρότασή μας έχουμε αξιολογήσει όλα τα υφιστάμενα στοιχεία που υπήρχαν και υπάρχει και μια πολύ λεπτομερής έκθεση του Κοινοβουλίου και όπως είπα τώρα ε, τα κράτη-μέλη θα αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των επιλογών της Τη ζώνη ώρα για να κάνουν μια επιλογή με αυτή τη βάση. Να περάσουμε στον τρίτο γύρο συζήτηση. Ναι, παρακαλώ, κύριε Γκρίφιν. Ε, με συγχωρείτε, Γερζή. Ε, δεν επανέρχομαι ο συνήθω, αλλά πραγματικά είστε πρόεδρος ε, που του μεταχειρίζεται όλου ισότιμα. Ε, α, με συγχωρείτε, εδώ πέρα έχω την αίσθηση ότι διαβάζει κάποιο σενάριο εκπρόσωπος της Κομισιόν και δεν ακούει το τι είπαν οι βουλευτές. Και ε, πραγματικά θα προτιμούσα μια απάντηση που θα λαμβάνει υπόψη τα όσα λέμε ως αιρετή εκπρόσωπη σε αυτήν την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Uh, thank you. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ ηγητά, σχεδόν λησμονήσαμε ότι σημαντικότερη ήταν η δική σας παρέμβαση για όλους μας. Ποια έποψη σε την όλη συζήτηση, πώς βλέπετε όλη αυτή τη συζήτηση που διεξήχθη στην Επιτροπή μας, συνεργασία, τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Ε, κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γνωρίζουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να συμβάσει ε, και να ακουστούν διαφορετικές απόψεις. Ε, προσπάθησα να σεβαστώ και τις δύο πλευρές ως ηγητής ε, και την πλευρά που λέει όπως και εγώ ότι είναι σημαντικό να καταργηθεί η αλλαγή της αλλά πρέπει να σεβαστούμε και την άλλη πλευρά που έχει επιχειρήματα και λέει είμαστε εναντίον. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για εμένα είναι να βρούμε μια λογική ε, οδό. Δηλαδή να πούμε ξεκάθαρα ε, αφενός ότι δεν θα γίνει αυτό εντός της προθεσμίας που προτείνει η Κομισιόν ε, και δεν είναι σωστό, είναι άσχημο για εμάς να βγαίνει ο πρόεδρος της Κομισιόν και να λέει θα το κάνουμε τώρα άμεσα. Γιατί μετά αυτό δημιουργεί προσδοκίες και εμείς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, κάποια πράγματα που πρέπει να δούμε και καλό θα ήταν να έχουμε μια αξιολόγηση από την Κομισιόν και είναι ξεκάθαρο και όλοι το ξέρουν ότι τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή έχουν πολύ δύσκολες συζητήσεις και δυσκολεύονται πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία Και βεβαίω, εντάξει, μπορεί και η Επιτροπή να πει, βεβαίω είναι μια γνωμοδότηση, να πει ότι εμεί αυτό θέλουμε, αλλά αυτό μετά απαιτεί τον χρόνο του και πρέπει να δούμε όλα τα πράγματα ε, στις λεπτομέρειες χωρίς, δεν έχει νόημα να λέμε υπέρ ή κατά χωρίς να μπούμε στην ουσία. Αναμένω λοιπόν τις επόμενες ημέρες κάποιες ενδιαφέρουσες ε, συζητήσεις με τους κοιόδης εισηγητές Υπάρχουν οι προθεσμίες, ε, τα έχουμε πει με τη γραμματεία. Υπάρχει κάποια πίεση χρόνου. Όπως σας είπα, εγώ θέλω να υπάρχει κάποιος ε, αμοιβαίος σεβασμός, ε, να ακουστούν οι διαφορετικές απόψεις και δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Θα υπάρξει μια ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιο πριν δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο πέρα από το ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Ωραία, ευχαριστώ. Έξοχα. Ο συνήθω ο εισηγητή τη ε, Επιτροπή ΙΤΡΕ είναι ανοιχτό σε όλε τι προτάσει και γνωρίζει ότι μέχρι την ψηφοφορία στην Επιτροπή ΙΤΡΕ δεν γνωρίζουμε τίποτα. Το αποτέλεσμα θα γνωστοποιηθεί τον Μάρτιο. 4 Μαρτίου η ψηφοφορία στην Καθήλια Αρμόδια στην Επιτροπή Μεταφορών 4 Μαρτίου, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών στην Επιτροπή Ήτρε, 30 Ιανουαρίου, την επόμενη εβδομάδα, θυμηθείτε την επόμενη εβδομάδα, 30 Ιανουαρίου, είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Σημαντικότατα αυτό για την έκθεση του συναδέλφου Σβέν Σούλτσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ καλή συζήτηση. Σημαντικότατο θέμα για όλους μας και για τους πολίτες μας μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο, το υπαριθμό 9. Την εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Νεολαία και με παρουσίαση να καλωσορίσω με μεγάλη μου χαρά με μεγάλη χαρά λέω Υποδεχόμαστε τρεις νέους για την εκδήλωση αυτή, για την νεολαία της Ευρώπης, για Τζόναθαν Κουκ, Φραντσέσκα Επίσκοπο και Φρόικε Γκέμπραου, που θα παρουσιάσουν ιδέες που ίσως να αφορούν το μελλοντικό έργο της Ήτρε και πιο συγκεκριμένα για την ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, οικολογικό σχεδιασμό, επιχειρηματικότητα και ε, έλεγχο του γονιδίου και επεμβάση στο γονίδιο. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τη ρομποτική. Λοιπόν, η επέμβαση στο γονίδιο και επιχειρηματικότητα που σας είπα. Να σας υπενθυμίσω σε όλους, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ότι αυτή η εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Νεολαία έραβε χώρα την 1η και 2η Ιουνίου 2018 στο Στρασβούργο. Συμμετείχαν πάνω από 9.000 νέοι. Συζήτησαν διάφορες ιδέες που αφορούσαν και το μέλλον της Ευρώπης και θα θέλαμε να παρουσιάσουμε κάποια αποτελέσματα των συζητήσεων που ακολούθησαν. Αν επιτρέπετε, θα ξεκινήσω με πρώτο μιλητή τον κύριο Τζόναθαν Πουκ, ο οποίος θα παρουσιάσει δύο ιδέες εν γέννη. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα θεμάτων. Την επέμβαση στο γονίδιο και παρακαλούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τον Τζόναθαν. Έχεις το λόγο, Τζόναθαν. Καλημέρα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ και μπορώ να παίξω ένα μικρό ρόλο στις συζητήσεις του Κοινοβουλίου. Είμαι πανεπιστημιακός ερευνητής και εξετάζω τα θέματα διοντολογία στη βιοτεχνολογία και ασχολούμαι με ε, τι επεμβάσει στα γονίδια διαφόρων οργανισμών. Το έθεσα θέμα συζητήσεω στην εκδήλωση που έγινε για την νεολαία, για την επανάσταση του DNA, όπω αποκαλείται. Θέλω να προτείνω δύο αλλαγέ που προτείνονται από την συζήτηση όσον αφορά τη σκόπιμη απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Οι τροποποίησει που πρότεινα θέλουν να εξασφαλίσουν ότι ταιριάζει καλύτερα ε, η οδηγία ε, στην απελευθέρωση διαφόρων ε, επεμβάσεων τροποποιημένων οργανισμών, φορέων διαφόρων μολύνσεων όπως είναι τα κουνούπια. Θα πρέπει η οδηγία γενετικά τροποποιημένου οργανισμού να τροποποιηθεί, ούτω ώστε να απαιτείται κάποια συνένεση, ούτω ώστε να γίνονται διάφορε δοκιμέ διαφορή ασθενειών που περιέχουν συνθετικά γονίδια. Λοιπόν, θα διευκρινίζουμε πώς υπάρχει διάδραση μεταξύ ε, κανονισμών και οδηγιών και δοκιμών και να υπάρχει ένα πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων και για συνεργασία μεταξύ των αξιωματούχων για τη δημόσια υγεία και εκπροσώπων των διαφόρων μελών τη κοινότητα που είναι στόχο. Το άρθρο 9 τη Οδηγία Γενετικά Τροπημένου Οργανισμού απαιτεί ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν διαβούλευση με το κοινό μετά την με απελευθέρωση γενετικά τροπημένων οργανισμών και θα πρέπει να δίνουν τι κατάλληλε πληροφορίε ε, γι' αυτό. Όμω υπάρχει και η άλλη άποψη ότι θα πρέπει το κοινό να έχει ε, μεγαλύτερη προστασία ηθική όσον αφορά τι δοκιμέ, όσον αφορά γενετικά τροποποιημένους φορεί ασθενειών. Γιατί, διότι τέτοιε δοκιμέ συμπεριλαμβάνουν διάφορα στοιχεία που αφορούν περιβαλλοντική ε, ε, πυροβολητικά πελάματα, αλλά και κλινικές δοκιμές και ίσως να χρησιμοποιούνται και διάφορα στοιχεία δεδομένα ατόμων. Ακόμα και αν αυτές οι δοκιμές η δημόσια υγεία θα είναι υποφελής για την δημόσια θα πρέπει να έχουμε αυστηρές, αυστηρά πλαίσια για την προστασία των κοινοτήτων. Όπω και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία έχει θέσει ένα πλαίσιο, λέει ότι επαρκή κανονισμοί σε αυτό το τομέα θα πρέπει ε, να επιβάλλουν και δημοκρατικέ διαδικασίε για να μπορεί το κοινό να συμμετέχει και να μπορεί να παρεμβαίνει στι όλε τι διαδικασίε. Αυτέ οι διαδικασίε θα ξεπερνούν την κοινότητα που θα είναι παθητικοί αποδέκτε αυτών των πληροφοριών. Οι αξιωματούχοι δημόσια υγεία θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων με εκπροσώπου τη κοινότητα και θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων. Οι δοκιμέ θα πρέπει να γίνουν ε, μετά από αυτή τη διαδικασία, αν τα μέλη της κοινότητας ε, το εγκρίνουν σύμφωνα με τις διάφορες πολιτικές διαδικασίες που προβλέπονται. Κάποιες αρχικές δοκιμές γενετικά τοποποιημένων φορέων ασθενειών εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως επεκρίθησαν διότι δεν εξασφάλιζαν επαρκή συμμετοχή και έγκριση κοινότητα. Σαν εκπρόσωπο των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να νομοθετεί και να εξασφαλίζει ότι δεν θα πρέπει να διαπράξει τέτοια σφάλματα σε ενδεχόμενε μελλοντικέ δοκιμέ. Δεύτερη σύσταση, είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει νομικά να θεσπίσει και να αναγνωρίσει συνεργάσιμο φορέα, όπου θα πρέπει να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας ε, Ασφαλείας Τροφίμων και της Υπηρεσίας για την πρόληψη και εξάλληψη ασθενειών, για να ε, μπορέσουν να δουν τι γίνεται όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα αυτά, του γενετικά τροποποιημένους φορείς ασθενειών. Λοιπόν, τι συζητήσαμε στην εκδήλωση. του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πιο λογικό και επιστημονικό όσον αφορά τι τεχνολογίε επέμβαση γενετική εν γέννη. Πιστεύω ότι αυτή η γενική ανησυχία που εκφράζουν οι νέοι εδράζεται επί του γεγονότο σε οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που διέπει γενετικά τροπημένου οργανισμού βασίζεται στην αρχή τη πρόληψη. Κάποιοι συμμετέχοντε ε, στην Ευρωπαϊκή αυτή εκδήλωση των νέων πιστεύουν ότι αυτή η αρχή ερμηνεύτηκε με έναν τρόπο ότι ίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει περισσότερο του κινδύνου των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών χωρί να εξετάζει τα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει από αυτού. Αυτό κάπου αλλού αναφέρθηκε και θα το επαναλάβω εδώ. Ανταυτού θα πρέπει να κάνω συγκεκριμένη σύσταση σχετικά πώ μπορεί να αυξηθεί η αυστηρότητα επιστημονική αξιολογήσεω των κινδύνων που απαιτείται στο συγκεκριμένο πλαίσιο των γενετικά τροποποιημένων φορέων ασθενειών στα πλαίσια τη οδηγία του 2001, γενετικά είναι οργανισμοί υπόκειται σε αξιολόγηση κινδύνου που γίνεται από την Υπηρεσία Ασφάλεια των Φήμων, την Ευρωπαϊκή. Όμω, πολλοί από του κινδύνου και τα ωφέλη τη τεχνολογία επέμβαση στα γονίδια ξεπερνούν το πεδίο εφαρμογή αυτή τη τεχνογνωσία του φορέα. Αυτό ο φορέα που προτείνει να δημιουργηθεί είναι απαραίτητο ώστε να αξιολογεί επαρκώ του διάφορου κινδύνου και τα ωφέλη που δημιουργούνται από την επέμβαση στα γονίδια. Επιδημιολογία, δημόσια υγεία και βιοπικιλότητα που λαμβάνονται υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ήδη έχει κάνει διάφορα δημοσιεύματα συνεργαζόμενοι με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και Έλεγχο των Ασθενειών κατά Καταπολέμηση άλλων βιολογικών κινδύνων, όπω ασθένειε που ε, ε, περνούν μέσω φορέων. Και αυτό ο φορέα προτείνω εγώ θα παρέχει ανεξάρτητη επιστημονική συμβουλή και ε, βοήθεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επίση, θα σε καλή θέση να αναθεωρεί τι κατευθύνε γραμμέ που υπάρχουν για αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων των γενικά τροπικών οργανισμών και πώ μπορούν να γίνουν διάφορε δοκιμέ βάσει αυτών των φορέων ασθενειών που έχουν υποστεί επέμβαση όσον αφορά τα γονίδια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε ένα πάγωμα, να παγώσουμε τι δοκιμέ. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθήσει τη σύμβαση του ΟΗΕ όσον αφορά τη βιολογική ποικιλομορφία και να μην ε, επιβάλλει αυτό το πάγο, αυτό το μαρατόριμο. Αυτό δεν απαιτείται από τη στιγμή που γίνεται σωστός, σωστή εξολόγηση κινδύνου που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο του κινδύνου που δημιουργούνται από τι νέε αναδυόμενε τεχνολογίε, αλλά και τη φύση του κόστου να διαλέξει κανεί να κρατήσει την καθιστική ατάξη. Κλείνοντα, όπως καταλαβαίνω εγώ, αυξάνεται αυτός ο τομέας και πρέπει να λάβουμε αποφάσεις για τους κινδύνους και τα ωφέλη των τεχνολογιών που έχουν βαθιά ε, επίδραση στην ανθρώπινη υγεία ενδεχομένω. Το Κοινοβούλιο τώρα θα πρέπει να δει κατά πόσο έχει τους ανδεχόμενους το επαρκής ε, φορεί που μπορούν να κάνουν την εξολόγηση των ωφελών και των κινδύνων που ε, απορρέουν από αυτέ τι νέε αναδυόμενε τεχνολογίε των γονιδίων. Ευχαριστώ, Τζόναθαν. Να πω μερικά λόγια. Να πω δύο λόγια. Είπε ότι είσαι 30 ετών, το έχω γράψει εδώ στο φακελό μου και είσαι Βρετανός και μεταδιδακτορικός ερευνητής που ασχολείται με την ηθική φιλοσοφία στο κέντρο της Οκφόρδης για την πρακτική ηθική. Και είσαι επικεφαλής ε, του project για ε, την ε, ηθική που έχει να κάνει με την διέγερση του εγκεφάλου. Πολύ εντυπωσιακό, έχεις δημοσιεύσει πάρα, πολλά άρθρα για την ε, γονιδιακή τροποποίηση στους ανθρώπους και στα ζώα και έχεις ε, γράψει στην εφημερίδα Guardian, ε, έχεις παρουσιαστεί στο BBC και στο Global News Network. Πάρα πολύ μεγάλη πείρα ως νέος επιστήμονας. Και τώρα το λόγο έχουν τα μέλη. Κυρία Γκρίφιν. Καλώς ορίσατε. Χαιρόμαστε που σας έχουμε και τους τρεις ε, εδώ. Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση, Τζόναθαν, και θα ήθελα να ρωτήσω τη γραμματεία. Θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε όλες ε, τις ε, παρουσιάσεις και των τριών, έτσι ώστε ε, όσοι δεν είναι σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο να μπορούν να εξετάσουν τις παρουσιάσεις και να δουν τι μπορούμε να προωθήσουμε. Αλλά, Τζόνι, νομίζω ότι ήσουν ε, και την ε, προ... στην προηγούμενη συζήτηση όταν πολλοί βουλευτές είπαν ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη και τις επιπτώσεις στην υγεία. Ένα μέρος του προβλήματος που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι έχουμε πάρα πολλές ε, τοποθεσίε υδραυλική ρογμάτωση ε, και αυτό λαμβάνει χώρα ενώ οι επιπτώσει στην υγεία και στο περιβάλλον του φράκινγκ της υδραυλική ροχμάτωσης δεν έχουν εξεταστεί πλήρω και είναι κρίμα γιατί οι πολίτε λένε ότι δεν θέλουμε να το έχουμε αυτό στην πίσω βλή μα, δεν ξέρουμε τι επιπτώσει για την υγεία μα και για τα παιδιά μα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι δεν γίνονται σεβαστέ ε, οι απόψει του και θα ήθελα να εξετάσει την νομοθεσία που ήδη ε, ψηφίσαμε. Όλα τα κόμματα συμφωνούσαν να βάλουμε τους πολίτες στο επίκεντρο ε, της νομοθεσίας για την καθαρή ενέργεια. Εμείς ε, θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι πρώτα θα βάλουμε τις θέσεις της ανάγκης των πολιτών. Και εμείς ζητήσαμε να μας αποδείξουν πώς ε, ε, λαμβάνουν ε, υπόψη και διαβουλεύονται τις τοπικές κοινότητες και τους νέους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να τυκμπόξουν να λένε το κάναμε αυτό. Θέλουμε πραγματικούς μηχανισμούς αποτελεσματικούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να γνωρίζουμε ποιες είναι οι απόψεις των πολιτών μας. Και όλες οι ιδέες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για, τον, για την νεολαία μπορούν ε, να μας βοηθήσουν και είναι ευπρόσδεκτες. Πρέπει να υπάρχει πραγματική διαβούλευση με την κοινότητα. Θα πρέπει να έχουμε μηχανισμού που να βοηθούν του ανθρώπου, ε, οι οποίοι κανονικά δεν έχουν φωνή, να μπορεί να ακουστεί η φωνή του σε ό,τι πλήττει το μέλλον του. Σα ευχαριστώ που είστε εδώ Βλέπετε ότι σημαίνουν διάφορα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ βέβαια ε, είμαι υπέρ του να ψηφίζουν οι πολίτες και να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Μαρτέν. Εγώ δεν ε, είμαι ειδικό στο θέμα αυτό, αλλά θέτεται μία ερώτηση, ένα θέμα που είναι εδώ και αφορά το θέμα της διαφάνειας και τα δημοκρατικά όργανα που μας ε, οδηγούν στο να αποφασίζουμε για τα θέματα αυτά. Και δείτε τι συμβαίνει τώρα με τη Μοσάντο και το Κλειφοσάτ. Δείτε τι γίνεται με την ΕΦΣΑ. Κατηγορούμε την ΕΦΣΑ ότι ουσιαστικά αντέγραψε μία έκθεση της Μοσάντο. Επομένως, το θέμα είναι τα λόμπι που κρύβεται από πίσω και προέρχεται από, προέρχεστε από την ε, πρωτεύουσα του λόμπι και είναι σαν τη χολυστερίνη. Υπάρχει καλό και κακό λόμπι. Όμως πρέπει να υπάρχει και μία αντιεξουσία μεταξύ, μέσα σε εισαγωγικά γιατί, κοιτάξτε, και εμείς ε, οι βουλευτές δεν είμαστε ειδικοί σε πολλά ζητήματα και πρέπει να έχουμε και ένα διαφορετικό βλέμμα και εσείς μας το προσφέρετε αυτό και στην αρχή της ε, θητείας θα ήθελα να έχω ακούσει την άποψή σας, ε, όχι μόνο γιατί είστε νέος, ε, αλλά και γιατί παρουσιάζετε μια άλλη κριτική άποψη. Εμείς θα πρέπει να έχουμε την υποχρέωση να αμφισβητούμε τη δημοκρατία, να, μάλλον να θέτουμε ερωτήσει σε σχέση με τα δημοκρατικά μα συστήματα και πώ η κοινωνία των πολιτών μπορεί να καταπολεμήσει τα λόμπι, Πώ πρέπει, πώς να βρούμε την κανονική ισορροπία. Σα ευχαριστώ λοιπόν για όλε τι διευκρινήσει που μα δώσατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σκόκλιτσεκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους που ασχολούνται με πρακτικά πράγματα. Ε, δεν είμαι σίγουρος εάν έχω καταλάβει ποιες είναι οι πρακτικές επιπτώσεις ε, των όσων λέγονται εδώ. Εγώ όμως είμαι τεχνικός ε, και αναζητώ τους στόχους των πραγμάτων. Εάν υπάρχει συζήτηση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, είναι διάφορα αν μιλάμε για ζώα ή φυτά ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να είμαστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτήν την συζήτηση. Κανείς μας δεν είναι ειδικό σε αυτόν τον τομέα. Εγώ ήμουν στον τομέα της οικοδομής, δεν είχα κάποια σχέση με αυτά τα θέματα, αλλά να σας πω το εξής. Με κάποιες αρρώστιες οι οποίες ε, υπάρχουν όταν υπάρχει μια αλλαγή των γονιδίων του ανθρώπου. Ε, μπορεί να εκδηλωθούν οι συνέπειες ε, μετά από δύο ή τρεις γενιές. Οπότε θα ήθελα να υπάρξει ένα πάνελ ειδικών για να λάβουμε τις πληροφορίες. Δεν είμαστε παντογνώστες, αλλά θα πρέπει να φτάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας πραγματικά σε βάθος. Γιατί καμιά φορά όταν μιλάμε για ζώντες οργανισμούς ε, και πολύ μικρές λεπτομέρειες παίζουν τεράστιο ρόλο. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Το έβλεπα αυτό στους ασθενείς του. Και συμφωνώ, πράγματι έχετε δίκιο. Πρέπει να εργαστούμε εδώ πέρα στην πρόταση αυτή με την Κομισιόν και μπορούν να το στηρίξουν πολλοί συναδελφοί μας. Αλλά είναι απολύτως απαραίτητο ναι, είναι πολύ προσεκτικές οι έρευνες αυτές τις αξιολογήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομα, Τζόναθαν, εάν μου επιτρέπετε, είπατε σωστά ότι βεβαίως ε, η κοινωνία δεν είναι απλά παθητικός δέκτης. Πώς βλέπετε την δικιά μας την επιρροή. Παράδειγμα του χάρη πώς θα μπορούσε να αλλάξει η επιρροή μας το χρονοδιάγραμμα ε, μιας ε, ε, κλινικής δοκιμής. Γιατί έχω και προσωπική εμπειρία. Γιατί δοκίμασαν επάνω μου μια πειραματική θεραπεία. Δεν ήταν εύκολο πριν από ένα χρόνο και ακόμα υποφέρω. Αλλά είναι αναγκαίο από καιρού καιρών να πάει κανεί στην κλινική και να πει ναι, συμφωνώ, εντάξει, δεν είναι πλήρως ε, ελεγμένο, αλλά δοκιμάστε το πάνω μου. Ε, Πώ το βλέπετε αυτό από σκοπιά ήθικης. And maybe GMO. GMO, you see. GMO. Ναι, και για του γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ναι, έχουμε του συναδέλφου εδώ από την Επιτροπή Περιβάλλοντο και Γεωργία που ενδιαφέρονται πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά κανόνα θέλει να προστατεύει τους πολίτες. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ε, είμαστε ανοιχτό μυαλί ως προς αυτό και αναφέρατε κάτι τέτοιο. Νομίζω. Ακόμα και αν θεωρούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προστατεύουμε τους πολίτες μας, δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να έχουμε πάντα την ίδια άποψη με τους πολίτες μας. Καμιά φορά πρέπει να πηγαίνουμε παραπέρα από τις σκέψεις και τις προσδοκίες των πολιτών μας. Α, συγγνώμη κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό ότι έρχονται οι νέοι να εκφραστούν εδώ και να μας διαβιβάσουν τις σκέψεις τους και το έργο τους. Όμως ας ε, μην γινόμαστε και ε, λαϊκιστές ε, και να λέμε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι καλό, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, ότι είναι καταστροφικό το λόμπι. Όχι, όλοι ασκούν πίεση και εγώ το ίδιο κάνω εντός της ομάδας μου. Όταν παίρνω το σχάρι είμαι εισηγήτρια για ένα σημαντικό θέμα και εγώ ασκώ πίεση, όλοι κάνουν λόμπι λοιπόν. Και δεν θα πρέπει να κάψουμε και τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Είναι σημαντική και άσκηση πίεσης γιατί μας επιτρέπει να τις ακούσουμε όλους. Αν ε, το ε, θεωρήσουμε ε, με έναν ε, τρόπο που είναι δηλαδή να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο να περισσότερες πληροφορίες από όλα τα μέρη και αν ε, οι βουλευτές έχουν την αίσθηση της ευθύνης και κάποια στιγμή κλείσουν την πόρτα και αρχίζουν να σκέφτονται και να προβληματίζονται για να προτείνουν την καλύτερη δυνατή λύση, τότε πολύ καλά. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Κοιτάξτε, με ενδιαφέρουν ε, πάρα πολύ τα θέματα της υγείας ε, και τα θέματα που αφορούν ε, την φαρμακοβιομηχανία και μπορώ να σας πω ότι εργάζομαι πολύ και με τις ενώσεις ασθενών, είναι απαραίτητες και δεν μπορούμε να εργαστούμε για θέματα υγείας χωρίς να έχουμε τις σχέσεις με τις ενώσεις ασθενών γιατί αυτές ε, μπορούν ε, πραγματικά να μας μεταδώσουν τι αισθάνονται οι ασθενείς αλλά και οι επαγγελματίες της υγείας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε έντιμοι και όλα αυτά να τα βλέπουμε από κάποια απόσταση και να προσέχουμε για να μην δελικοποιούμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε, Τζόναθαν. Πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας ε, και για τη συμμετοχή σας στο θέμα αυτό. Ίσως θα μπορούσα να ξεκινήσω με τη δική σας ερώτηση για το ποια είναι η διαφορά από μια ε, κλινική ε, δοκιμή για ένα άτομο. Νομίζω ότι όταν ε, συμμετέχει ένα άτομο θα πρέπει ε, ο ασθενής να δώσει τη συνένεσή του, θα πρέπει να συμφωνήσει για να συμμετέχει σε αυτή την κλινική δοκιμή. Όταν μιλάμε όμως ε, για δοκιμές στη δημόσια υγεία, όταν ε, μιλάμε παραδείγματο χάρη για την απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων κουνουπιών, ε, δεν είναι δυνατόν να ρωτήσει κάθε έναν άνθρωπο στην κοινωνία αν δέχεται να δεχτεί, να υποστεί του κινδύνου έναντι των ωφελών. Έτσι λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η σωστή δημοκρατική διαδικασία και νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε για να το δούμε αυτό σε διάφορα εθνικά πλαίσια. Επίσης, ε, έχει να κάνει και με το σχόλιο που έκανε η βουλευτής ε, για τις ενώσεις ασθενών. Μπορούμε να σκεφτούμε και τις ομάδες ενός ασθενών. Εγώ ε, μιλώ ουσιαστικά για κλινικέ δοκιμέ, ε, προληπτικών φαρμάκων, Επομένω, όλος ο πληθυσμό ε, θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει ασθενή. Έτσι λοιπόν όλο αυτό αποτελεί μια πραγματική δημοκρατική πρόκληση. Και κάποια άλλα σημαντικά σημεία. Ναι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη χρήση αυτή τη τεχνολογία. Αυτό με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο με το κύριο που το ανέφερε, όμως ε, θα πρέπει να δούμε πώς αξιολογούμε και τους κινδύνους και τα ωφέλη της τεχνολογίας. Μπορεί εύκολα να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια νέα τεχνολογία, να υποθέσουμε ότι πρόκειται για μια νέα τεχνολογία και επομένω θα πρέπει να υιοθετήσουμε την αρχή της προφύλαξης και να θέσουμε μορατόριου, αλλά Μπορεί να μιλάμε και για μια περίπτωση που μπορούσαμε να έχουμε μια τεχνολογία που θα μπορούσε ε, σοβαρά ε, να μειώσει την, ε, τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβαστές. Παραδείγματος χάρη, είχαμε 20.000 θανάτους από ελαιονοσία και βέβαια είναι εκτός της Ευρώπης, αλλά το 2014 το ECDC σε μία έκθεσή του είπε ότι θα αυξηθεί ο κίνδυνο ζωσιμάτων που μεταδίδεται με διαβαστέ στην Ευρώπη λόγω τη κλιματική αλλαγή. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να συζητούμε τώρα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας για την υδραυλική ρογμάτωση, όμως είναι παρόμοια η κατάσταση όπου έχουμε μία ευρεία παρέμβαση στην κοινωνία και πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δημοκρατικές διαδικασίες και να υπάρχει συμφωνία των πολιτών για μία ενδυνάμει επικίνδυνη επέμβαση. Ε, και νομίζω ότι πρέπει να πάμε περαιτέρω από το απλώς να ενημερώνονται οι πολίτες και να παρουσιάζουμε την επέμβαση αυτή ως κάτι ε, Θα πρέπει να υπάρχει μία συμμετοχική διαδικασία, αλλά το πώς θα το οργανώσουμε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το απαντήσουμε τα επόμενα έτη. Σας ευχαριστώ πολύ, Τζόναθαν, για την παρουσίασή σου και για τις ε, προτάσεις σου και φυσικά που σε τις ε, ερωτήσεις. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια, την ε, Φραντσέσικα Επίσκοπο. Όποτε φαίνεται όλο και πιο νέοι είναι οι ομιλητές εδώ. Είστε Ιταλίδα εκπροσωπείτε την Ιταλία και έχετε πτυχίο αστυνομική από το Πανεπιστήμιο της Πίσα και από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τώρα δραστηριοποιείστε στο Πανεπιστήμιο της Πίσα και είστε και ερευνήτρια στην ανώτερη σχολή Σαντάνα και υλοποιείται διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα για τα είναι ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την προστασία των δεδομένων και την αποδοχή των χρηστών της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη δική μας Επιτροπή, γιατί έχουμε και μια έκθεση τη πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη στην Επιτροπή αυτή και ψηφίσαμε πριν από ένα μήνα την έκθεση αυτή και τώρα ε, συζητούμε το πρόγραμμα της ψηφιακής Ευρώπης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη επταετία, γιατί θα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα καινούριο πρόγραμμα, το πρόγραμμα της ψηφιακής Ευρώπης και εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Μιλάμε πιθανότητα για 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλα αυτά τα θέματα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα στα μέλη της Επιτροπής. Είμαι Φρανσέσκα Πίσκοπο και χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω δύο ιδέες που επεξεργαστήκαμε στην εκδήλωση στα πάνελ της Ευρωπαϊκής Νεολαία για τη ρομποτική και την για τεχνητή νοημοσύνη. Η πρώτη ιδέα είναι να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική. Ε, χρειάζεται έλεγχο αυτών των δύο τομέων. Είναι τεράστια πρόκληση για την Ευρώπη. Έλλειψη, καθυστέρηση, ανεπάρκεια ε, ρύθμιση ίσω επιτρέψει τεχνολογίε οι να δημιουργηθούν που δεν σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχέ ή να έχουν ανατριχιαστικές, ε, να έχουν μάλλον να παγώσουν την εξέλιξη τεχνολογία και καινοτομία. Σαν ερευνήτρια πολύ συχνά βλέπω την κατάσταση όπου ρυθμιστική και ρυθμιστικά εμπόδια εμποδίζουν επιχειρήσεις και πανεπιστήμια να αναπτύξουν ε, προϊόντα και να προωθήσουν την έρευνα. Για να υπάρξει σωστή διαχείριση του θέματος, προτείνω η Ευρώπη να δημιουργήσει λοιπόν έναν φορέα για τη ρομποτική και τεχνική νομοσύνη, εκτελεστικό φορέα με ίδια χρηματοδότηση με τρεις λειτουργίες που θα αναλάβει. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προσφέρει ε, σε ευρωπαϊκού και εθνικού φορεί, τεχνογνωσία επιστημονική και τεχνολογική και να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ θεσμών και ενδιαφερομένων κύκλων και να προωθεί πρωτοβουλίε για την πρόθεση της ρομποτική και τη χρήση αυτή. Δεύτερον, να αναπτύξει και να επιβάλλει και να επικαιροποιεί συνεχώ κανόνε για τον έλεγχο, οι δοκιμέ για την πιστοποίηση και τυποποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών εφαρμογών και τέλο, εξίσου σημαντικό, θα πρέπει να διαχειρίζεται διοικητικά μέτρα όπως μητρό για συγκεκριμένες εφαρμογές ρομποτικής, ταμεία για αποζημίωση και να μπορούν να κατατίθενται οι βέλτιστες πρακτικές και να λαμβάνονται υπόψη για τις δοκιμές και επιστοπίσεις νέων προϊόντων. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί φορέζητη ρομποτική. Είναι κάτι που συστήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα χρησιμοποιούσε άλλε πρωτοβουλίε για την κατεύθυνση των δράσεων Ευρωπαϊκής Ενώσης, όπως συζητήσει σε ομάδες εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικού φορεί υψηλού επίπεδου. Και αυτό έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πριν κάποιε εβδομάδε είχαμε το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τη δεντολογία, για τεχνητή νοημοσύνη, που ήταν το αποτέλεσμα εργασιών τη ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου για τεχνητή νοημοσύνη. Παρά τη σημασία αυτών, αυτά τα εργαλεία δεν έρουν την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή υπηρεσία τη ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη. Διότι αυτός ο παρέχει τεχνογνωσία και θα έχει και λειτουργίες ρυθμιστικές και, κανονι... και διοικητικές ε, σε επίπεδο οριζόντιο και διοργανικό. Και αυτή είναι η μόνη λύση που μπορεί να εξασφαλίσει έγκαιρη, πλήρη συντονισμένη αποτελεσματική προσέγγιση ρυθμιστική και έτσι η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί στον τομέα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης και θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές της Ευρωπαϊκής και έτσι οι πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν από την ψηφιακή επανάσταση. Ζητώ από εσά, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ήτρε, να ζητήσετε να δημιουργηθεί ε, μια τέτοια ευρωπαϊκή υπηρεσία για τη ρομποτική και για την τεχνητή ε, νοημοσύνη. Δεύτερη ιδέα που έχω και θα ήθελα να συζητήσουμε είναι να απτυχθεί Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Εξολογήσεως της Ρομποτικής. Η ρομποτική τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν εξαιοπρέπεια την ιδιωτικότητα, την αυτονομία και την ασφάλεια των ανθρώπων σε ψυχικό και φυσικό επίπεδο και δημιουργούνται νομικά θέματα και διοντολογικά. Από τη μία πλευρά, η καινοτόμα φύση τέτοιων συσκευών μαζί με μακροπρόθεσμα απρόβλεπτες συνέπειες της χρήσης δυσχεραίνουν την, να εντοπίσουν οι ερευνητέ και επιχειρήσει και να αξιολογήσουν του κινδύνους που ίσω να δημιουργηθούν και να του μειώσουν του κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, οι νομοθέτε και εκείνοι που διαμορφώνουν την πολιτική έχουν ανεπαρκή στοιχεία για να καθορίσουν κατά πόσο οι συσκευέ που δημιουργούνται είναι νόμιμε για να ρυθμίζουν από ιδέα μέχρι παραγωγή του προϊόντος τη διαδικασία και εποπτεία της αγοράς και να αξιολογούν πόσο αποτελεσματικά και αποδοτικά είναι τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί μέσω νομοθεσίας. Γι' αυτό προτείνω η Ευρώπη ενδεχομένω μέσω τη προτεμένη υπηρεσία για τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική και με τη βοήθεια εμπεριγνωμόνων από διάφορου τομεί, μήπω θα έπρεπε να δημιουργήσει ένα μηχανισμό αξιολογήσεω τη χρήση τη ρομποτική, ένα μέσο να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσει που ασχολούνται με τη ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη και θα πρέπει να κοινοποιούν το πώς συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις. Αυτός ο μηχανισμός θα αντικαταστήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται αντιμετώπιση κινδύνων, όπως είναι η προστασία των δεδομένων. Και θα πρέπει σε ένα ενιαίο εγγραφό να συλλέγονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον αντίκτυπο και τις μειώσεις, μηχανισμό μείωσης της κινδύνους. Ε, που μπορεί να δημιουργηθούν από τη χρήση διαφόρων αυτονόμων οχημάτων και ρομπότ και αυτό να γίνει στα διάφορα στάδια εξέλιξης. Σε μία άνωθεν προσέγγιση, η αξιολόγηση κινδύνων θα βοηθήσει αυτούς που χωρούνται με τη ρομποτική να αναλύσουν τους κινδύνους και να τους μειώνουν τους κινδύνους που ίσως να προκύπτουν από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Αυτό είναι κάτι που συνάδει με υπάρχουσες προδιαγραφές και δημιουργούνται νέες κατευθυντήρες γραμμές και βαθμολόγηση, άμα χρειάζεται. Σε μια κάτωθεν προσέγγιση μπορούμε, ε, μπορούν οι ρυθμιστές να εντοπίσουν κενά ρυθμιστικά και να συλλέγουν στοιχεία για το είδος των κινδύνων που δημιουργούνται από διάφορες κατηγορίες ρομπότ και τέλος, εξίσου σημαντικό, θα υπάρχει μια βάση για υστέρων νομοθετική αξιολόγηση που μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση και επικαιροποίηση του υφισταμένου νομικού πλαισίου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Φραντσέσκα. Και τώρα θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Καταρχήν ο κύριος Ζωρίνιο έχει το λόγο. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Φραντσέσκα, για τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδέες που μοιράστηκε μαζί μας. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ε, για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ τα ζητήματα που έθεσες και εσύ. Στο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη έχουμε συμπεριλάβει και ιδίω στα κεφάλαια που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την αναγκαιότητα να υπάρξει μια ηθική αξιολόγηση, δηλαδή να υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας ε, που θα τηρείται σε όλα τα προγράμματα που θα εγκριθούν και θα εφαρμοστούν. Όμως, ε, όπως σίγουρα γνωρίζετε, η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση είναι το κλειδί και θέλουμε να ξέρουμε αν η τεχνολογία θα εξυπηρετήσει τους ανθρώπους ή, ή αν θα είναι οι άνθρωποι που θα υπηρετήσουν τελικά την τεχνολογία. Κυρίως ε, όταν ε, μιλάμε με τους νέους, εγώ συνομιλώ πάρα πολύ και με τους μαθητές μου γιατί διδάσκω στον τομέα αυτό ε, βλέπουμε ότι έχουμε κάποιους ε, ευφυείς αλγόριθμους που θα βρίσκονται στη βάση όλων αυτών ε, και όλοι, μαζί αν δεν εφαρμόσουμε τις βελτίστες πρακτικές, αν δεν έχουμε ορθές αξίες, αν δεν κατορθήσουμε να είμαστε ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τη μηχανή, τότε η μηχανή θα απορροφήσει το δικό μας μοντέλο ε, λειτουργία στην κοινωνία και θα βελτιώσει την κοινωνία μας. Όμως αν αντιθέτως, αν ε, έχουμε εγωιστικές πρακτικές, ε, αν χάσουμε τον έλεγχο της τεχνολογίας, αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να έχουμε κάποια θέμητα πλεονεκτήματα πάνω στους ομοίους μας, τότε θα δημιουργήσουμε μια ψηφιακή κοινωνία όπου όλα τα κακά θα πολλαπλασιαστούν. Δηλαδή θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ανισότητες ε, και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και γι' αυτό ο προβληματισμός που μας κατέθεσε εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, το θέμα της υπηρεσίας, του φορέα. Ε, Εμεί η ψηφιακή Ευρώπη δημιουργούμε 28 κόμβους. Έχουμε αρχίσει ε, να σκεφτόμαστε για να έχουμε μια πιο συνεκτική Ευρώπη ότι σε μια νέα ψηφιακή κοινωνία ένας φορέας, ένας οργανισμός δεν θα πρέπει να είναι ένα νέο υλικό κέντρο αλλά θα μπορούσε να αποτελεί ένα δίκτυο ικανοτήτων. Τελειώνω Πρόεδρε. Και σε σχέση με τη δεύτερη ερώτηση, την αξιολόγηση αντικτύπου, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η αξιολόγηση αντικτύπου, αλλά θα πρέπει Συγγνώμη, συνάδελφε, έχω επτά συναδέλφους στον κατάλογο. Ναι, ναι, το ξέρω, Πρόεδρε, ότι εσείς χειρίζεστε πολύ δίκαια το χρόνο. Απλώς ήθελα να απαντήσω στο δεύτερο θέμα για την αξιολόγηση κινδύνου. Έχουμε δύο σενάρια πάντοτε. Το σενάριο σχετικά με το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος, αν έχουμε μια θετική εφετηρία και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αν έχουμε μια αρνητική βάση αξιών για αυτή τη δυναμική. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχουμε και άλλη μια νεαρή ενώπιόν μας και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σας παρακαλώ, έχω έξι άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο για να θέσουν ερωτήσεις στη Φρατσέσκα. Παρακαλώ να μην μακρηγορήσετε. Λυπάμαι γι' αυτό. Ο Λόπες Βερβάνιο, παρακαλώ. Η κυρία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικές οι παρουσιάσεις σας. Οι δύο που ακούσαμε και σίγουρα θα είναι και η τρίτη. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ε, συμφωνώ απόλυτα με τη σαφήνεια των όσων παρουσιάσετε και φυσικά από ό,τι φαίνεται έχει υπάρξει και πολύ μεγάλη έρευνα εις βάθος όλα τα θέματα της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης ε, αποτελούν ε, πολύ σημαντικά θέματα για μας. Εγώ συμφωνώ με την αναγκαιότητα να ιδρυθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός πέρα από τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν από την πλευρά των χωρών αλλά όπως είπε και η ομιλήτρια, νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια Ευρώπη που θα συγκλίνει περισσότερο και με μεγαλύτερη συνοχή και νομίζω σε αυτό συμβάλλουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Βλέπουμε ότι λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί σε άλλου τομεί και είναι πολύ καλό εργαλείο. Επίση, πρέπει να έχουμε και ένα μηχανισμό αξιολόγηση αντικτύπου. Συμφωνώ με αυτό συμφωνώ σε σχέση με την προστασία των δεδομένων και τα στοιχεία που παρουσιάσατε. Όμως θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε και μια αξιολόγηση αντικτύπου για το ε, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος, η συνέπεια στην αγορά εργασίας, γιατί βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας επανάστασης και αν εμείς ε, θέλουμε να έχουμε μια υπεύθυνη ανταγωνιστικότητα, πρέπει να ξέρουμε ποιος θα είναι και ο αντίκτυπος ε, στους εργαζομένους. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, γιατί σίγουρα χρειάζεται ένα στοιχείο κλειδί για τη ρομποτική που είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών. Και η εμπιστοσύνη αυτή μπορεί να κερδιθεί μόνο αν ε, είμαστε διαφανείς και μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά περί διαφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Κόχλιτσεκ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Βασικός ε, κανόνας της ρομποτικής είναι ότι τα ρομπότ δεν θα πρέπει να βλάπτουν τον άνθρωπο. είναι ένα βασικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε γιατί εισάγουμε όλο και περισσότερα ρομπότ και κάποια από αυτά είναι αυτορυθμιζόμενα. Ποιος είναι υπεύθυνο λοιπόν αν γίνει κάποιο λάθος από αυτά τα ρομπότ. Τρίτον, πρέπει να προωθήσουμε τη ρομποτική, ναι, αλλά όσον αφορά τώρα την υπηρεσία εγώ θα προτιμούσα κάποιον και μηχανισμό αξιολόγησης αντικτύπων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Γιατί είναι τόσο πολλά τα ζητήματα έτσι ώστε μια υπηρεσία που θα βρίσκεται σε ένα σημείο, Βρυξέλλες ή αλλού, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Πατρίτσια Τόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι κάθε φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κάθε δύο χρόνια, εγώ βλέπω ότι είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι, πολύ όριμοι και πολύ ικανοί. Θα ήθελα να σταθώ όσο είπα η Φραντσέσκα Επίσκοπο, γιατί είναι θέματα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε εμείς. Και από τις πολλές προτάσεις μας έδωσες θα αναφερθώ σε δύο. Το πρώτο αναφορά το μηχανισμό αξιολόγησης ε, των κινδύνων. Ε, νομίζω ότι είναι μια ιδέα που θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή και ε, ε Έδωσε ε, και κάποια στοιχεία για τις ηθητικές ε, πτυχές ε, και δεν είναι ποτέ τέλειο αυτό, αλλά είναι απόλυτη ανάγκη και μπορούμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ρομποτική. μπορούμε να έχουμε μια στρογγυλή τράπεζα για το θέμα αυτό, όμως άλλοι που εργάζονται αλλού στη Σιγκαπούρη έχουν τελείως διαφορετική στάση έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πτυχή που είναι νομική πτυχή αλλά αφορά και τη φιλοσοφία και το δίκαιο. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Εμείς ε, πάλι ε, υπό μια νομική σκοπιά φτάσαμε σχεδόν να πούμε ότι υπάρχει σχεδόν νομική προσωπικότητα του ρομπότ και ε, ίσως ε, είναι υπερβολικό αυτό, είπε το Κοινοβούλιο. Όμως ε, το να έχουν νομική ευθύνη η παραγωγή, παραδείγματος χάρη το ρομπότ, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ αν και στη χώρα μου, όταν δεν ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα, λέμε να φτιάξουμε ένα οργανισμό και μετά βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους που είναι στη δημόσια διοίκηση να είναι σε αυτόν τον οργανισμό. Γιατί να μην αξιοποιήσουμε τις ικανότητες, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο, παραδείγματος χάρη, και όχι πάντοτε να να αναθέτουμε τις αρμοδιότητες σε εξωτερικά υποκείμενα. Εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Διοίκηση έχει τις απαραίτητες ε, ικανότητες ε, ε, και να μην προσφεύγουμε σε εξωτερικούς όπως πάντοτε. Σας ευχαριστώ κύριο Σταμπουράνο. Ευχαριστώ. Παιδιά, θα απαντήσω και στους δυο σας. Να πω κάτι που καμιά φορά ξεφεύγει αλλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχει σύγκληση μεταξύ βιοτεχνολογιών και ψηφιακών τεχνολογιών. Έχουμε τέτοια πρόοδο όσον αφορά την τεχνολογία την ψηφιακή, που σήμερα και στο μέλλον περισσότερο θα μπορούν να μιμιστούν τους βιολογικούς αλγορίθμους. Οπότε τίθεται το θέμα αυτό που συζητείτε σε διάφορα περιβάλλοντα και στο Κοινοβούλιο, που ίσως πρέπει να μπει περισσότερο στην ημερήσια διάταξη Δηλαδή ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουμε πάνω σε αυτά. Καλό να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε κινούμενοι θεμάτων φιλοσοφικών και βιοπολιτικής, διότι τεχνική και επιστήμη οδηγούν σε πολλά πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Αλλά χρειάζεται να αποφασίσουμε ποια κατεύθυνση θα πάρουμε. Ποια είναι αυτά που μπορούν να γίνουν και ποια αυτά που δεν πρέπει να γίνουν βάσει φιλοσοφίας και βιοηθικής αν θέλετε και σε ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου ευτυχώς ακόμα έχουμε ευαισθησία ανθρωπιστική και δοντολογική ανώτερη, δόξα τω Θεώ, από τις άσπρες του κόσμου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την τεχνολογική ανάπτυξη χωρίς όρια και χωρίς ε, κανόνες, όπως τις είπα και στην Κίνα, όπου ήδη ε, γίνεται γενετική, γενετικός πειραματισμός και να ακολουθήσουμε έτσι απλά αυτούς, διότι υπάρχει κέρδος και που οι άλλοι μπορούν να προχωρήσουν πιο πέρα από εμάς. Λοιπόν, το θέμα είναι αν θέλουμε να παρεύουμε στη γενετική κληρονομιά των φυτών, των ζώων και των ανθρωπίνων όντων και να, κρύ... και να προσωμιώσουμε την ευφυΐα και τεχνητά και τις βιολογικές λειτουργίες. Δεν πλέον τεχνικό πρόβλημα, διότι προχωράει η τεχνολογία και δείχνει και θα δείξει ότι μπορεί να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά είναι ένα θέμα βιοπολιτικής και ηθικής. Ευπρόσδεκτοι οι ερευνητές που ασχολούνται με τη φιλοσοφία, διότι ίσως την πολιτική είναι στιγμή να σκέφτεται περισσότερο φιλοσοφικά από ό,τι τεχνολογικά και περισσότερο ανθρωπιστικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Βυρκούνεν είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστήσω και εγώ τους νεαρούς ερευνητές που ήρθαν σήμερα να μας παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είμαστε Επιτροπή Έρευνας και βιομηχανία. Θέλουμε να ακούσουμε τι ιδέε των νέων ερευνητών για το τι πρέπει να γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο και όταν μιλάμε για ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα τα τελευταία χρόνια και στην Επιτροπή μας και στο ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί όταν μιλάμε για την ψηφιοποίηση τα ρομπότ γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη είναι μια κατακαιρματισμένη αγορά γιατί υπάρχει διαφορετική νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Και τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει 30 διαφορετικά νομοθετήματα για να μην υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των κρατών μελών και να υπάρχει μία ενιαία ψηφιακή αγορά. Και έχουμε αποφασίσει για όλες αυτές τις ε, πρωτοβουλίες. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για μία ενιαία ψηφιακή αγορά. Βέβαια, τώρα έχουμε νέες προκλήσεις, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία από αυτές, μεταμορφώνει έτσι την κοινωνία μας και βλέπουμε και σε παγκόσμια κλίμακα. Στη ΣΥΠΑ ή στην Κίνα επενδύουν τρει και πέντε φορές περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη και για να είμαστε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να επενδύουμε πολύ περισσότερο στην έρευνα και στην καινοτομία. Και όπως είπατε, Φραντσέσκα, πέρσι η Κομισιόν συνέστησε αυτήν την ε, ομάδα και βεβαίως έχουμε και την ηθική πτυχή και έχουμε και διαφορετικές αξίες ίσως στην Ευρώπη από ότι οι ανταγωνιστές μας ε, και μιλάμε ακριβώς για την ηθική της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ε, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά όπως είπε και η συνάδελφος, η Πατρίτσια, αυτή είναι η καλύτερη λύση. Ε, εντάξει, τώρα δεν ξέρω για να συστήσουμε μια νέα υπηρεσία, γιατί συχνά αυτό ακούμε, ότι χρειάζεται μια νέα υπηρεσία να το αναλάβει και μετά δεν θα έχει πόρους. Ε, αν δεν έχει πόρους μετά δεν θα βοηθήσει κτλ. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συντονιστούμε επαρκώς. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, λυπάμαι συνάδελφοι, δεν έχουμε χρόνο για συζήτηση. Ε, συναρπαστικά όλα αυτά τα οποία λέμε. Ε, Φραντσέσκα, ήρθε η ώρα να κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά σας. Το να απαντήσω σε δύο λεπτά είναι πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσω να το απαντήσω όλα μαζί. Η αφετηρία είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπατε πολλοί από εσάς, ότι δηλαδή η Ευρώπη χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και πρέπει ακριβώς να δούμε και την ανακοίνωση της ε, Κομισιόν πέρσι που έχει αυτόν ακριβώς τον στόχο. Πρέπει λοιπόν να βασιζόμαστε σε δύο αρχές. Η πρώτη είναι να κάνουμε επιλογές ε, όχι μόνο με βάση το τι είναι τεχνικά εφικτό αλλά και τι μορφή θέλουμε να έχει η τεχνολογία για να προωθήσουμε τις αρχές μας. Ε, και να ε, εργαστεί η τεχνολογία για εμάς. Και το άλλο είναι ακριβώς η ανάγκη να υπάρξουν αυτές οι στοιχείες της δεοντολογίας ευρία ταινία, δηλαδή τι αντίκτυπο έχουν και στην κοινωνία τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το άλλο στοιχείο που θεωρώ απαραίτητο είναι αυτό ε, της σωστής ρύθμισης ε, και ακριβώ ε, εγώ ανέφερα την πιθανότητα δημιουργίας μιας υπηρεσίας για να δημιουργηθούν κάποια στοιχεία ακριβώς συνεργατικής διοίκησης που θεωρώ ότι θα μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα από έναν φορέα που θα έχει έναν ρόλο ε, ουσιαστικότερο από συμβουλευτικό που έχουν άλλοι φορείς. Και καταλήγοντας εδώ, θα έλεγα ότι η ιδέα μιας υπηρεσίας δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι Μιλάμε μόνο για ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι θα είναι πιο αποτελεσματική σε ένα δίκτυο και με τους εθνικούς φορείς και υπ' αυτήν την έννοια θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς για όλες τις σχετικές επιχειρήσεις που εργάζονται πάνω στο θέμα και τώρα ακριβώς προσπαθούμε να δούμε με μεγάλη δυσκολία τους πολλούς και διάφορους κανονισμούς που ισχύουν γύρω από το θέμα. Τέλος, η ανάγκη να δούμε ποιος είναι υπεύθυνο για την τεχνολογία και την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι σαφές ότι δεν έχουμε αυτή την στιγμή κάποιες λύσεις ε, για τα θέματα αυτά ε, για κάποια λύση ρομποτικής ή τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι υπεύθυνη γιατί όσες ικανότητες και αν έχουν είναι ε, μηχανήματα τα οποία δεν είναι ε, υποκείμενα με ηθική και ο άνθρωπος πίσω από αυτά αποφασίζει. Οπότε θα πρέπει ακριβώς ε, να υπάρχουν οι σωστές ηθικές αρχές για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών και να υπάρξουν και κάποιοι κανόνες εξάντε και το ποιος επίσης ε, θα είναι υπεύθυνο ε, εκ των υστέρων εάν υπάρξει ένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ για τις Ευχαριστώ λοιπόν για τα σχόλια, για τους φορείς, για τις υπηρεσίες. Έχουν πολλές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα οι υπηρεσίες όπως προτείνεις ε, είναι απαραίτητες και η Επιτροπή Ήτρε θα το εξετάσει. Πάμε στο τελευταίο μιλήτη. Την κυρία Γκεράου που είναι Γερμανίδα, μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη, νότια του Βερολίνου. Μετά το γυμνάσιο, ένα χρόνο έκανε θελοντική δουλειά στο Ινστιτούτο για την έρευνα της Βαλτικής, στο Ροστόκ. Μετά από αυτό, από επιστήμες πήγαινε στη μηχανολογία και αποφάσισε να ασχοληθεί με τεχνολογία βιογενετικών πόρων και από το βιογραφικό σας βλέπω ότι θέλετε να συνδυάζετε τεχνολογία με οικολογικές απόψεις και ασχολείστε ε, και είστε στη ΜΚΟ, οι νέοι φίλοι της φύσεως της Γερμανίας από το δημοτικό δηλαδή είσαστε σχεδόν εκεί, από πολύ μικρή. Έχετε λοιπόν το λόγο. Καταρχάς, εκτιμώ το ότι είμαι εδώ και έτσι μου δίνεται την εντύπωση ότι με έχει πλησιάσει πολύ η Ευρώπη. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ και που ε, μου διαθέτετε χρόνο και με ακούτε. Πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει ένα κανονισμό για το σχεδιασμό ηλεκτρικών συσκευών σε τμήματα μπορούν να επισκευάζονται πολύ καλά και έτσι ένα κομμάτι, ας πούμε, της εικόνα, κομμάτι που, της εικόνας μπορεί να αλλάζεται εύκολα. Λοιπόν, χρειάζεται να αλλάξουμε ε, τη ζωή μας για να αντιμετωπίσουμε αλλαγή του κλίματος και θα πρέπει να θέλουν οι πολιτικοί να πετύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από είναι τεχνητά Κάθε δύο χρόνια αλλάζουν περισσότερο κινητό τηλέφωνο τους, παρόλο που λειτουργούν και βλέπω πολλού που έχουν στην καθημερινή ζωή του σπασμένη οθόνη διότι η επισκευή κοστίζει πολύ, χρειάζεται χρόνο και δεν μπορεί να το επισκευάσει κανεί μόνο του. Οπότε θεωρούμε τελικά ότι καλύτερο είναι να πετάμε κάτι να διορθώνουμε. Με αυτή το σχεδιασμό σε τμήματα, μια σπασμένη κάμερα μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιον και το υπόλοιπο τηλέφωνο που χρησιμοποιείται για περισσότερο χρόνο. Έτσι και άρα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ακόμα και οι του τεχνικού υλικού μπορεί να α, γίνεται. Δεν χρειάζεται να πάει σε ένα καινούριο τηλέφωνο, λειτουργεί καλύτερα μέσα επικαιροποίηση. Αυτό ισχύει για ταμπλέτε και για τα τηλέφωνα που πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν ηλεκτρονικέ μηχανισμού ανάγνωση και άλλε συσκευέ μπορούν μπορεί να γίνονται έτσι. Θα πρέπει να καθοριστούν πρότυπα που για τα πια ε, ανταλλακτικά μπορούν να αλλάζονται. Και εγώ προτείνω ε, καλάχιστα. Η εικόνα, η μπαταρία, η κάμερα, ξεχωριστά, η μνήμη, η εξωτερική θήκη, τα κουμπιά και οι θύρε ε, επίσης και εκεί που είναι το σύστημα αποστολής και λήψης, λοιπόν τα διάφορα κομμάτια θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για παραγγελία μέσω του ίντερνετ. Εγώ πιστεύω ότι θέλουν οι άνθρωποι να αγοράζουν βιώσιμα προϊόντα αν είναι εφικτό και η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας. Το βλέπετε και στην έκθεση ε, που έχει δημοσιευτεί. Γι' αυτό στην, ε, είχαμε από τις ιδέες ήταν αριστή ιδέα μου. Στις μελέτες μου έμαθα ότι ένα κίνητρο για τον μηχανικό χρησιμοποιεί την ενέργεια και τις διάφορες πηγές αποδοτικά. Και το θέμα της βιωσιμότητας πολύ συχνά το συζητούν οι ερευνητέ και οι μηχανικοί. Όμως πολλά που είναι τεχνικά εφικτά μπλοκάρονται από τους οικονομολόγους που θέλουν να συνεχίσουν το επιχειρηματικό μοντέλο και θέλουν να έχουν οικονομία κλίμακας. Μόνο χρειάζεται πολιτική δράση για αλλαγές Λοιπόν, όταν έκανα έρευνα, είδα, βρήκα δύο μικρές επιχειρήσεις που είχαν φτιάξει κινητά τηλέφωνα με κομμάτια ανταλλάξιμα. Και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Για τι μεγάλε βιομηχανίε η βιωσιμότητα δεν είναι ακόμα θέμα που του απασχολεί. Ο κόσμο θέλει μια καλή ηλεκτρονική συσκευή. Όσον αφορά τι τεχνικέ δυνατότητε, βλέπουν. Αγοράζουν αυτό που έχει καλύτερε επιδόσει παρόλο που θα μπορούσαν να αγοράσουν ένα τηλέφωνο πιο βιώσιμο. Άρα η αγορά πρέπει να τροποποιηθεί. Οι ευρωβουλευτέ μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξουν την αγορά, να διαμορφώσουν το μέλο τη ηλεκτρονική παραγωγή. Δεύτερη ιδέα. Μικρά προσαρχικού κεφαλαίου να δώσουν σε πολλά προγράμματα που χρησιμοποιείται τεχνολογία για ε, δραστηριότητα επιχειρηματική φιλική προς το περιβάλλον και να μπορούμε να κινηθούμε και μέσω τοπικής υποδομής για βιώσιμο κόσμο και καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο, ε, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Αλλά δεν έχουμε κάνει μεγάλε αλλαγέ παρόλο που τελειώνει ο χρόνο. Αντί να δίνουμε μεγάλε χορηγίε σε μεγάλε επιχειρήσει, μήπω ήταν αποτελεσματικότερο να δίνουμε σε μικρότερα ποσά ποσών σε πολλού ανθρώπου να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν μια, μια νοοτροπία φιλική προ το περιβάλλον. Χρειάζεται εκδημοκρατισμό των μέσων, των τεχνολογιών, των δεξιοτήτων για καλύτερε λύσει και τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίζει από εκεί και πέρα τι πιο βιώσιμε, Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογία θα πρέπει να συναθρίζει την έρευνα και την τεχνολογία. Έχουμε και ένα πρόγραμμα στη Γερμανία, το Exist, που το προσπαθεί να το κάνει αυτό. Αυτοί οι μαθητέ οι μητέρε στο σπίτι, αποκλείονται και αυτοί με τεχνική κατάρτιση. Και η ανεργία επίση των νέων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά από το πρόγραμμα. Άρα, πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να παράξουμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και γρήγορα και να ενθαρρύνουμε όσο δυνατόν περισσότερους ε, τις ιδέες τους να τις κάνουν επιχείρηση και προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει συνεργαστεί κατά άποψή μου με φυστάμενες δομές ανοιχτών εργαστηρίων, εργαστηρίων, χώρους hackers. Και υπάρχουν σε κάθε χώρα αυτοί οι φορεί και υπάρχουν υποδομέ που πολύ συχνά βρίσκεται σε εταιρείε και ερευνητικά ιδρύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που να μπορεί να βοηθήσει κάποιου να ξεκινήσουν στι τοπικέ κοινότητε. Μέσω του προγράμματο να επιδοτούνται εργαστήρια, να διδάσκονται άνθρωποι που χρησιμοποιούν μηχανήματα και πώ η πτυχή τη βιωσιμότητα επηρεάζει τα προϊόντα και την κατασκευή των προϊόντων. Έτσι μπορούν πολλοί να μάθουν, πολλοί που έχουν κίνητρο και θέλουν να κάνουν κάτι. Άρα εδώ έχουμε έφορο έδαφο για καλή διαφήμιση υπέρ τη βιώσιμη προσέγγιση. Χρειάζεται ενεργοποίηση των μικρών επιχειρήσεων και χρειάζεται στήριξη στην αρχική φάση. Παραδείγματο, ε, ε, ε, ξεκίνησε κάποιο το καθαρισμό και αν όχι, ήθελε να, να δημιουργήσει επιχείρηση, αλλά να στηριοποιηθεί. Τώρα έχει μεγαλώσει, έχει γίνει επιχείρηση και απασχολεί πάνω από 80 ανθρώπου που καθαρίζουν ωκεανού. Κάθε ιδέα μπορεί να λυθεί. Έχει κίνητα αυτό που θέλει να κινηθεί να βρει λύση για τη βιωσιμότητα και αν στηριχθεί μπορεί να βοηθήσει. Χίλια ευρώ μπορεί να δίνονται στην αρχή το αίτημα να, η αίτηση πρέπει να είναι ε, απλή και θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κριτήρια της χάρτας για βιωσιμότητα του ΙΕ για να υπάρχει σωστή επιλεξιμότητα για τα χρήματα. Μπορεί να, να διαφημιστεί και αυτό. Χρειάζονται χρήματα για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα. Μετά καθοδήγηση από τοπικό δίκτυο. Λοιπόν, προτείνω στα μέλη της Επιτροπής Ήτρε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα για να δημιουργήσετε τοπικά εργαστήρια και να χρηματοδοτούνται μέσω μικρών χρηματοδοτήσεων σε μικρά ποσά οι τοπικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή, πολύ καλή πρόταση. Εμείς στην Επιτροπή Ήτρε είμαστε υπεύθυνοι για πολλά, πολλά σημαντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάδελφοι, ποιος θα ήθελε το λόγο. Ο κύριος Κόχλιτσεκ, καταρχήν. Ε, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε μια 23 χρόνια σε ποια νεολαία ήσασταν. Α, των ε, φίλων της ε, φύσης. Ναι, έχω καλές σχέσεις με αυτή την οργάνωση. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσω τσεχικά. Αν και ίσως θα ήταν καλύτερο να μιλήσω γερμανικά στην ε, νεαρή κυρία, αλλά εντάξει, δεν Λοιπόν, έχω τρει ερωτήσει. Κοιτάξτε, αυτός ο τρόπος προσέγγισης, ο σταδιακό υπάρχει ήδη σε ε, πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες ακριβώς για να μπορούν τα κομμάτια μιας συσκευή να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα. Ε, δηλαδή λέτε αυτό το οποίο ήδη λένε κάποια έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό Έχουμε παραδείγματο χάρη σήμερα ενιαίου φορτιστέ, ενιαίε μπαταρίε, Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση και μπορώ να την υποστηρίξω. Το δεύτερο για τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις είπατε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν ε, δραστηριότητες. Δεν ξέρω πώς έχουν τα πράγματα σε άλλες χώρες, αλλά στην ε, Τσεχία έχουμε έτσι σε αυτές ε, θερμοκοιτίδες για τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις ε, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες υπηρεσίες εκεί πέρα, βοήθεια με τα λογιστικά κτλ. Λοιπόν, και είναι περιορισμένη διάρκεια. Είτε μετά τα πάνε καλά, και φεύγουν από τη φωλιά ας πούμε ή αλλιώς ε, ατύχησαν. Αλλά έτσι γίνεται και μετά. Οι νέοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι με την ε, τεχνολογία πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να το κάνουν αυτό και στα σχολεία έχουμε εταιρείες οι οποίες κάνουν εικονικές ξεναγήσεις, έχουμε το Εράσμους ακριβώς για την επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά οι ιδέες σας και θα τις στηρίξω. Σας ευχαριστώ. Ο συναλφός Ταμπουρανό, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, πραγματικά συγκινήθηκα από τον ενθουσιασμό που βλέπω σε μία νέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ για την αναγκαιότητα τα ηλεκτρονικά προϊόντα να αποτελούνται από δομοστοιχεία, γιατί επικεντρωνόμαστε κυρίως ε, στην ομοθεσία, στην δυνατότητα ανακύκλωσή τους, ε, ε, όμως εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια αμερικανική μάρκα που είναι πάρα πολύ λειτουργική, αλλά τελικά μου έσπασε ένα τμήμα και ε, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω την ε, μπαταρία που ε, τελικά συνέχιζε να λειτουργεί. Εγώ θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από τους επιχειρηματίες υπάρχει πολύ μεγάλη αντίσταση απέναντι σε αυτή την ιδέα. Τώρα, το Κοινοβούλιο πολλές ε, φορές έχει κάνει προτάσεις υπέρ της βιωσιμότητας, όμως το Συμβούλιο υποστηρίζει τα βιομηχανικά συμφέροντα και δυστυχώς ε, μπλοκάρει πάρα πολλές από τις ε, πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε εμείς εδώ. Σε ό,τι αφορά τώρα την μικρή χρηματοδότηση, ναι, θα έπρεπε να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες σε μία σειρά ανθρώπων που έχουν ε, δημιουργικές ιδέες. Ίσως ε, να είναι λίγα τα χίλια ευρώ, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δίνουμε κάποια μικρά ποσά, ε, κυρίως τώρα που βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη και στην Ιταλία λείπει εντελώς ιδέα μιας νέας μορφής παιδείας για την ψηφιακή μετάβαση και φυσικά θα ξεκινήσει από ανθρώπου που μπορεί να είναι σήμερα παιδιά ή έφηβοι, αλλά τουλάχιστον στην Ιταλία, όπω και σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, δεν υπάρχει μια νέα διδακτική, μια νέα μοντοσοριανή μέθοδο που να μπορεί να προετοιμάσει του ανθρώπου για την ψηφιακή μετάβαση και να κάνει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ε, σε τι βρίσκονται ενώπιον όταν βάζουν τα στοιχεία του ε, στα δίκτυα κοινωνική δικτύωση ε, και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν στην καθημερινή ζωή και την παρουσία της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Η κυρία Λόπες, παρακαλώ, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Εγώ πιστεύω ότι η πρότασή σας ε, για, τα... Ε, για το σχεδιασμό ε, βάση δομοστοιχείων ε, θα συνεισέφερε από το στοίχημα που έχουμε θέσει και εμείς εδώ στην Επιτροπή και αφορά την κυκλική οικονομία, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, μείωση της ε, ε, κατανάλωσης και αυτό συνάδει με την ε, πρόταση αυτή. Όπως είπαν ε, και κάποιοι συνάδελφοι, πράγματι το Κοινοβούλιο σε αυτά τα θέματα συνεχίζει συνηθίζει να είναι πολύ πιο μπροστά από την ίδια την Επιτροπή και τα κράτη και επίσης συμφωνώ ότι θα πρέπει να δίνουμε κονδύλια για τέτοια project και αυτό έχει επίπτωση στο να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο κόσμο. Έτσι λοιπόν, το να αξιολογήσουμε και όλες αυτές τις περιβαλλοντικές πτυχές ε, θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την απόκτηση των κονδυλίων για να χρηματοδοτήσουμε τα καινοτόμα προγράμματα που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να σταλώ στο λόγο. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι. Να προσθέσω, αγαπητή Φράου, και ότι εμείς ως Επιτροπή είμαστε υπευθυνοί για τη βιομηχανία, την έρευνα, την ενέργεια, το ψηφιακό θεματολόγιο, την επιχειρηματικότητα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη διαστημική πολιτική, όλα αυτά μας απασχολούν σε αυτή την Επιτροπή. Είμαστε υπευθυνοί επίσης για το πρόγραμμα Horizon 2020 80 δισεκατομμύρια ευρώ, αρκετά μεγάλο ποσό και για άλλα προγράμματα όπως το COSME για τις ε, μικρές και μεσές επιχειρήσεις, τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά και για ένα νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, για τις ε, ψηφιακές δεξιότητες. Φυσικά είναι δυνατό να προτείνουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα όπως αναφέρατε εσείς, υπό την ε, ομπρέλα των πιλωτικών project. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσει να το λάβει υπόψη και η γραμματεία μας στην Επιτροπή Ήτρα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα δύο προγράμματα. Όμως, από τη δική σα σκοπιά, η καλύτερη δυνατή λύση θα ήταν εντός του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο Έρευνας. Ε, αυτό εντάσσεται στο πρόγραμμα Horizon 2020 στο επόμενο Horizon Ευρώπη. Το ορίζοντα 2020 είναι το πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 8, ενώ ορίζον Ευρώπη θα είναι το υπαριθμόν 9. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει πολλά κονδύλια για τους νέους επιστήμονες ε, για μεμονωμένα project, έργα των νέων επιστημόνων. Μπορείτε να το ελέγξετε και ε, θα δείτε εκεί ε, τα διάφορα προγράμματα, το Horizon Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε τις ιδέες σας. Να σας δώσω και τώρα το λόγο για τις τελευταίες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει μόνο οι ερευνητές να εφευρίσκουν κάποια πράγματα τα οποία θα είναι βιώσιμα, αλλά και άτομα με τεχνική εκπαίδευση και το σχολείο. Αλλά το σχολείο δεν θα πρέπει να δάσκει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί συνήθως ε, στο σχολείο είναι βαρετά τα πράγματα. Όμως ε, σε ένα εργαστήριο με τρισδιάστατους ε, εκτυπωτές, με ελεγχόμενα πράγματα που μπορεί κανείς να κάνει μια, μηχανήματα μπορεί να κάνει μια συγκόλληση ενός ε, τυπωμένου κυκλώματος. Αυτά παρέχουν κίνητρο. Κάποιοι, κάποιος είπε ότι ακριβώς ε, ο σχεδιασμός αυτός με εναλλασσόμενα εξαρτήματα υπάρχει σε κάποιους κανονισμούς. Δεν μπορώ όμως να αλλάξω την μπαταρία του κινητού μου. Ίσως θα μπορούσατε να πιέσετε τις εταιρείε να ακολουθήσουν αυτούς τους ε, κανόνες. Τώρα, είπατε ότι θέλετε να βελτιώσετε την κυκλική οικονομία. Θα ήθελα να επιμείνω στο ότι πρέπει να υπάρξει ένας κατάλογος και το πρώτο πράγμα στον κατάλογο αυτών είναι να αποφεύγονται τα σκουπίδια να υπάρχει επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και μετά να γίνεται ανακύκλωση ενέργειας με καύση και η τελευταία λύση να πετάγονται. Αλλά ακόμα και η ανακύκλωση είναι δύσκολη. Ξέρετε, δηλαδή το να βγουν τα τσίπ από διάφορα μηχανήματα. Είναι δύσκολο, χρειάζεται ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να αποφευχθεί η δημιουργία των σκουπιδιών και να τα ξαναχρησιμοποιούμε όσο περισσότερο γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις παρατηρήσεις σας αγαπητοί φίλοι. Είναι ε, μια πολύ ε, καλή δυνατότητα για όλους μας στην Επιτροπή μας. Είμαστε συνεχώς στο διαδίκτυο όλα όσα κάνουμε εδώ, όλα αυτά τα οποία λέμε. Να πω λοιπόν για τα ζητήματα διοντολογίας. Το λέει ο Τζόναθαν. Τα ζητήματα τέχνητης νοημοσύνης. Θα επηρεάσουν ε, ακόμα και την δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, το μέλλον ε, των οικονομιών μας. Και βεβαίως τα ζητήματα οικολογικής τεχνολογίας πώς θα αποφύγουμε την ρήπανση, τη βλάβη του πλανήτη. Όλα αυτά έχουν κρίσιμη σημασία και σας ευχαριστώ που ήρθατε και εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαία στην Περσινή και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε το εξαιρετικό σας έργο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον. Okay shaking. Go to the next point in our agenda. Πάμε στο επόμενο σημείο στην ημερησία μας διάταξη. Το υπαριθμόν 10. Αποστολή στην ε, αποκεντρωμένη υπηρεσία στην Πράγα τον Σεπτέμβριο του 2018. Επικεφαλής ήταν ο κύριος Μασιμίλιανο Σαλίνη, επικεφαλής τριών συναδέλφων. Στόχο είχε ακριβώς να δει το τι κάνει η υπηρεσία αυτή, ειδικά όσον αφορά το νομοθετικό έργο για το διαστημικό πρόγραμμα και τον ναι. ορίζοντα Ευρώπη. Μασιμιλιάνο, για πες μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα είμαι λακωνικότατος. Η αντιπροσωπεία πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα σπουδής και βάθυνση στο θέμα. Πριν ξεκινήσει η διαπραγματεύσεις είχαμε θέσει ένα στόχο Είχαμε, το μέσο της διαμόρφωσης συμβαστικών στο Κοινοβούλιο όταν κάναμε την αποστολή. Οπότε μπορέσαμε τελικά να ενισχύσουμε και τη διαπραγματευτική μας ε, ικανότητα μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Ε, και με πολύ ισχυρή εντολή πάω στον τριμερή διάλογο. θέση ισχύω. Δύο μέρες εργασιών είχαμε. Την πρώτη μέρα έγινε παρουσίαση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, πώς λειτουργεί, έγινε αναφορά συγκεκριμένα στα προγράμματα στο Έγνος και στο Γαλιλαίος, Είδαμε και ποιο είναι ο αντίκτυπο ο βιομηχανικό των συστημάτων μα του δορυφορική πλοήγηση. Διεξήχθη συζήτηση μεταξύ βουλευτών Ήτρε και της υπηρεσία με το διευθυντή και τους συνεργάτε τους. Αναλύσαμε όλα τα θέματα. Αυτά που αφορούσαν τον αντίκτυπο των αποφάσεων της Επιτροπής μας επί των δραστηριοτήτων της ε, υπηρεσίας. Κάποια συγκεκριμένα σημεία αναφέρθηκαν όπως ο ρόλος της υπηρεσίας σαν αρμόδια αρχή για ρυθμιζόμενες ε, κοινοφιλείς υπηρεσίες. Ε, ενδελεχέστατα συζητήσαμε το θέμα της ασφάλειας. Της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και ασφαλείας από πλευράς ε, ασφαλείας των προγραμμάτων Έγνους και Γαλιλαίος που αφορούν και το Security Accreditation Board, τη δουλειά που κάνει αυτό σοφορέας και που έχει αντίκτυπο και στις αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουμε για τα παραδοσιακά προγράμματα, όπως είναι ο Γαλιλαίος. Δεύτερη μέρα, μέσω ανταλλαγής απόψεων και μαρτυριών, ήρθαν σε επαφή με τους επιχειρηματίες και είδαμε διάφορες εφαρμογές του Γαλιλαίους και Έγνους. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Στο τέλος, μετά τη συζήτηση δεύτερης ημέρας, εστιαστήκαμε επί του περιεχομένου του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ποια είναι η δυνατότητα σύμπραξης μεταξύ προγραμμάτων του διαστημικού προγράμματος Space Program και του Horizon Europe και Invest EU και των άλλων προγραμμάτων που επηρεάζουν τη διαστημική μας στατηγική. Δύο μέρες πολύ σημαντικές, ε, πάρα πολύ χρήσιμες συζητήσεις και ωφελήθηκα και επίσης και για τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφε. Θα ήθελα να σας... Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω. Να ρωτήσω αν ο Εύζεν του Ζενόφσκι έχει να προσθέσει κάτι, γιατί ήταν και αυτός εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπε ο συνάδελφος. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Πραγματικά ήταν την κατάλληλη στιγμή. Ελάβαμε πολλές ε, πληροφορίες ε, σε σχέση με την ε, νομοθεσία η οποία είναι υπό κατάρτιση. Ως κάποιος ο οποίος πηγαίνει για δεύτερη φορά σε μια τέτοια ε, επίσκεψη. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν ε, η πρόοδος που έχει σημειωθεί εκεί πέρα. Ε, για μεγάλα βήματα. Είχαμε την πρώτη του συστήματος του δορυφορικού και εντωμεταξύ έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδο. Είμαστε στη φάση της εφαρμογή ξεκινούν νέα έργα τα οποία ήδη λειτουργούν, είναι συνδεδεμένα με άλλα έργα με τη σειρά του, ε, τα οποία επίσης λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, συμφωνώ με τον συνάδελφο, δηλαδή αποδείχτηκε πόσο σημαντικό είναι να δούμε κάποιες ε, απόψεις ε, παραδείγματος χάνει για τις διαδικασίες επιλογής και τα σχετικά για να μην έχουμε ασάφειες. Και είναι πάρα πολύ θετικό το να ξεκαθαρίζουν αυτά τα πράγματα. Επίσης συμφωνήσαμε στο ότι καθώς ε, υπάρχουν ε, νέες αρμοδιότητες, ε, διαβουλευόμαστε για αυτές, μιλάμε για αυτές και θα πρέπει να ενισχυθεί ταυτόχρονα και ο αριθμός των εργαζομένων για να ενισχυθεί ακριβώς η υπηρεσία αυτή και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι προστάτευσε επίσης ε, και τα θέματα προσωπικών δεδομένων και νομίζω αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το ποια προσέγγιση είναι απαραίτητη. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη, χρήσιμη για την προετοιμασία της ε, τρέχουσας ε, νομοθεσίας. Είναι λοιπόν μια υπηρεσία η οποία έχει καταφέρει να εκπληρώσει την αποστολή της. Τώρα πρέπει να γίνει το δεύτερο βήμα να συνεχιστούν αυτές οι δραστηριότητες ε, γιατί είναι ένα από τα πιο ακριβά έργα που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ήδη επιτυχημένο και από οικονομική σκοπιά και η περαιτέρω πρόοδο βεβαίω θα εξαρτηθεί από την συνολική εικόνα. Ο εισηγητή είναι ο συνάδελφο ο κύριο Σαλίνη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή αποστολή λοιπόν, λάβαμε πάρα πολλέ ε, πληροφορίε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι συμφωνούν λοιπόν ότι ήταν επιτυχημένη η αποστολή. Κύριε Κόχλιτσεκ, να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ χάρηκα ιδιαίτερος για το ότι έμειναν ικανοποιημένοι οι συνάδελφοι. Εγώ υποστηρίζω αυτή την υπηρεσία από την αρχή. Ήμουν αυτός που έλεγα πρέπει να πάει στην Πράγα. Ε, ακούω τώρα ότι λύθηκαν κάποια πράγματα και καλό είναι να έχει και περισσότερο προσωπικό και θεωρώ συμφωνούμε εδώ πέρα πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Σαλίνη θέλει να μας πει κάτι ακόμα. Οι παρατηρήσεις των συναδέλφων με βρίσκουν σύμφωνο και εμείς εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι το πιο λεπτό ε, τμήμα τη δέσμη μέτρων για το διάστημα αυτό που αφορά τις σχέσεις μεταξύ αυτού του οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εμβρήμης. Πρώτον ήταν αυτό. Δεύτερο, η σχέση αυτού του οργανισμού και του ESA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματο. Δηλαδή, το πακέτο που αφορά τη διακυβέρνηση θα είναι αυτό που θα συζητήσουμε περισσότερο, όμω η προπόθεση ε, συγγνώμη, μου φαίνεται ότι η εισαγωγή που έγινε με τον πρώτο τριμερή είναι εξαιρετική, γιατί και τα τρία θεσμικά όργανα είναι στο ίδιο μήκο κύματο και έχουν τον ίδιο στόχο. Το μόνο πρόβλημα προκαλείται από την ε, εντολή στο Συμβούλιο και να πω ότι είναι κάπως ε, ευάλωτη, εύθραστη η εντολή του Συμβουλίου, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές παρενθέσεις. Αν θα ξενήξουν αυτές οι παρενθέσεις, εντό Φεβρουαρίου θα κλείσουμε το δεύτερο τριμερή διάλογο και κατόπιν ε, θα συζητήσουμε και το θέμα των αριθμητικών στοιχείων στο πολιτές πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σαλίνη που ήταν ο επικεφαλής αυτής της ε, αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε σε δύο ώρες. Η Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Έχουμε ε, συνεδριάσεις με τους υπουργούς της Ρουμανίας ε, και κατόπιν ε, θα συζητήσουμε το θέμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Θα τα ξαναπούμε εδώ στις 2.30.